Bien, je vous prie de gagner votre place et j'ouvre la séance. Une séance. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Η συνεδρίασή μας στην ουσία θα είναι η συνεδρίαση της πρώτης ομάδας παρακολούθησης των διαδικασιών για την αναθεώρηση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου 14-20. Υπάρχουν κάποια σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να πω ότι μέσω γραπτής διαδικασίας έχουμε ένα αίτημα συνεργασίας από πλευράς της ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Ταμείο Αλληλεγγύης γύρω τώρα από τα πρακτικά της 19ης Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο, εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια. Τα πρακτικά όσα έχουν γίνονται δεκτά. Περνάμε λοιπόν αμέσως στη συνεδρίαση αυτής της ομάδας παρακολούθησης ή συνοδείας αν θέλετε, monitoring εν πάση περιπτώσει, Θέλω να σας καλωσορίσω όλους όσοι ήρθατε εδώ και ιδιαίτερα τους εισηγητές μας, τον κύριο Όλμπριχ και την κυρία Τομά, όπως και τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τα μέλη των Επιτροπών Ήτρε, Κοντ, που παίρνουν μέρος λόγω θέματος στη συνεδρίασή μας. Να καλωσορίσω επίσης και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις Γενικές Διευθύνσεις Προϋπολογισμού, RTB, Growth και Employ. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους επίσης για την παρουσία τους εδώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, έγινε μία συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς 1420 ξεκίνησε η συζήτηση επί τη βάση ενός εξαιρετικού εγγράφου το οποίο προετοίμασαν οι εισηγητές Τόμα και Ολμπριχτ. Όπως λέγεται στο έγγραφο αυτό, στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών η Επιτροπή Προϋπολογισμών θέλει να επανεξετάσει την λειτουργία και την εφαρμογή των νέων μέσων που προβλέπονται στα, στα μέσα, στα εργαλεία του νέου δημοσιονομικού επιδιώκοντας την επίτευξη της πολιτικής Ευρώπη 2020. Μας ανησυχεί επίσης η εξέλιξη του προϋπολογισμού. Υπάρχει μια δυσκολία να λάβουμε υπόψη μας κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ε, διαφανεί λόγω της κρίσης, κρίσης δημοσίου χρέους, κρίσης ελληνικής, και βλέπουμε να δημιουργούνται κάποιοι δημοσιονομικοί δορυφόροι ε, υπό τον τύπο καταπιστεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί ένα κατανοητό σημείο εξήγησης της λειτουργίας του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον μέσο πολίτη. Για να οργανώσουμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προετοιμασία της αναθεώρησης αυτής μέχρι τον Μάρτιο του 2016 θα έχουμε κάποιες ε, συνεδριάσεις σαν και αυτήν εδώ σήμερα. Αυτή η πρώτη ομάδα λοιπόν εποπτείας, αν θέλετε, ή παρακολούθησης ε, ασχολείται με τα βέσα ευελιξίας του πολιετούς δημοσιονομικού και για το θέμα των πληρωμών. Έχουμε ένα ραντεβού με τις πληρωμές. Τρία τμήματα, κάθε τμήμα με έναν ή δύο μιλητές και στο τέλος κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα καταθέσουν οι εισηγητές. Έχουν προετοιμαστεί και κάποια στοιχεία στο διαδίκτυο και θεματολογικά και γενικά Υπάρχει επίσης και ένα σημείωμα της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για τα θέματα των πληρωμών και τα έκτακτα μέσα. Θα πρέπει να κλείσουμε στις 11, γιατί στις 11 θα ψηφίσουμε. Και θα είμαι δυσάρεστος, δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, το να ε, συμπεριφερθώ με πολύ αυστηρό τρόπο σε σχέση με το χρόνο ομιλίας. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Όλμπρεχτ για πέντε λεπτά, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι, τα σχετικά δηλαδή με τα μέσα ευελιξίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του πολιετούς 14-20. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ήδη ως εισηγητές είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της παλιάς κατάστασης σήμερα. Να δούμε τι έγινε δηλαδή με την κατάσταση αυτή μέχρι τώρα και να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία έχει σαν στόχο όχι απλά να επανεξετάσει αλλά να αναθεωρήσει το επόμενο πι δελτα πι. Η αναθεώρηση του κανονισμού λοιπόν είναι ένα πράγμα. Για να αναλάβουμε όμως την ευθύνη αυτή οφείλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πι δελτα λειτουργεί. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της εισαγωγής των μέτρων ευελιξίας στα πλαίσια ε, του προγράμματος 15-20. Ε, μετά από δύο ήδη έτη λειτουργίας του νέου αυτού δημοσιονομικού πλαισίου, ε, το ερώτημα για να το πω απλά είναι δουλεύει το σύστημα ή όχι. Ε, υπάρχει η ευελιξία που απαιτείται ή όχι. Στο τέλος η ερώτηση θα τεθεί πιο σύνθετα. Απαιτείται περαιτέρω ευελιξία για το δεύτερο ε, τμήμα του πλαισίου αυτού του πολιετούς. Αλλά η πρώτη ερώτηση είναι να διαπιστώσουμε την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα στον τομέα της ευελιξίας. Για να το δούμε αυτό έχει σημασία να κατανοήσουμε την περιπλοκότητα των μέσων αυτών, διότι είναι υψίστως τεχνικά και περίπλοκα δομημένα. Η δεύτερη στρογγύλη τράπεζα ακριβώς αυτό θα προσπαθήσει να κάνει, το που βρισκόμαστε δηλαδή στην παρούσα φάση μετά τη χρήση των προβλέψεων ευελιξίας ε, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς έχει η κατάσταση σήμερα, ποιες είναι οι συνέπειες χρήσης ακριβώς αυτών των κανόνων ευελιξίας για το δεύτερο τμήμα, ποιες θα είναι μάλλον, του ε, ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η συζήτηση λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των προβλέψεων ευελιξίας, των ρητρών ευελιξίας, πώς έχουν πάει μέχρι τώρα τα πράγματα, τι πρέπει να αλλάξει από εδώ και πέρα και τι θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο. Ευχαριστώ κύριε Όλμπριχτ για την παρουσίασή σας και για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, γιατί για αναθεώρηση μιλάμε και όχι μια απλή επανεξέταση. Η πρώτη, αν θέλετε ο πρώτος γύρος των συζητήσεων είναι τα μέσα ευελιξίας. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε σωστά την αναφορά της ε, συζήτησής μας, θα δώσω τον λόγο στον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Επιτροπής. Έχετε για 15 λεπτά το λόγο κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Σιτά, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας ε, πρόσκληση. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάλυση που κάνατε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20. και με τα μέσα ευελιξίας ε, βουτάμε στα βαθιά ε, σε ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την ανάλυση. Νέα συζήτηση φυσικά δεν είναι νέο θέμα διότι τα περί δημοσιονομικού πλαισίου χρησιμεύουν στο, στον περιορισμό της ευελίξιας, ορίζοντας ανώτατα ωραία για βασικές κατα, κατηγορίες δαπανών για τις δεσμεύσεις αλλά και για τις πληρωμές για σειρά ετών και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποσκοπεί στον περιορισμό ακριβώς της ευελίξιας. Από την άλλη πλευρά, μέσα σε αυτό το περιοριστικό πλαίσιο μπορούμε να συμφωνήσουμε πολιετή προγράμματα χρηματοδότησης και μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσω πρόθεσμα την ε, χρηματοδότηση. Υπάρχει δηλαδή ε, μια ισορροπία σε κάθε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ανάμεσα στην ε, πειθαρχία και την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης αφενός και την ευελιξία αφετέρου. Πάντως, σε αυτό το πολιτές σε δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο δηλαδή, 2014 έως 2020, Έχουμε ξεκινήσει ήδη αργά, ε, με δύσκολα, ως προς την ευελιξία, ήδη από την αρχή. Θα ήθελα να σας θυμίσω τις διαπραγματεύσεις που μας οδήγησαν στο τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2013 μπόρεσε να εγκρίνει για πρώτη φορά ένα πολιετές πλαίσιο που σε πραγματικούς όρους ήταν μικρότερο από το προηγούμενο. Και υπήρχε μια ουσιαστικότατη διαφορά στο σύνολο των πιστώσεων ε, υποχρεώσεων και πληρωμών. Ε, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς ε, καμία δυνατότητα ε, παρερμηνίας, ξεκαθάρισε στις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών ότι δεν θα είναι βιώσιμο το πολιτές πλαίσιο αν δεν υπάρχει επαρκής ευελιξία. Η δέσμευση ως προς τη μέγιστη δυνατή ευελιξία που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα εκείνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήταν δίκαιο όμως να πω ότι είναι μας περιμένει ανηφόρα ε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδωσε ύψιστη προτεραιότητα σε αυτή την ευελιξία και με ε, στένος αγωνίστηκε για αυτή την ευελιξία. Αν δεν είχε γίνει αυτό από πλευρά του Κοινοβουλίου, δεν θα είχε προβλεφθεί αυτή η ευελιξία στο τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα είχαμε και τα ε, ρηξικέλευτα αυτά στοιχεία ευελιξίας ε, που μπορούμε και πάλι να τα αποδώσουμε στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν το ε, αποτέλεσμα για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 έως 20 που είπα είναι ούτως ή άλλως ε, περιοριστικό. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά και κάποια μέσα ευελιξίας που θα πρέπει να αναλύσουμε αναλύοντας αυτή τους την πτυχή, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξέλθει για αυτή την ε, πολιτική περίοδο. Θα ήθελα να κάνω εξ αρχής ένα βασικό διαχωρισμό θα αναλύσω τα μέσα ευελιξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία κατάρτισης κυλοποίηση του προϋπολογισμού. Δηλαδή όλα αυτά που θα αναφέρω μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Δημοσιονομική Αρχή για τον προϋπολογισμό και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό προς αποφάσεις που λαμβάνονται στο Συμβούλιο. Ε, έχουμε την ειδική ε, στο Συμβούλιο η ειδική πλειοψηφία άλλαξε και για τα ανώτατα όρια χρειάζεται τώρα ομοφωνία με σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το ευρύτατο μέσο ευελιξίας ε, είναι η ίδια η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η αναθεώρηση υπήρχε εξ αρχής ε, από την ίδρυση ε, του δημοσιονομικού πλαισίου, από τη θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου μπορούσαμε να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε τα ανώτατα όρια, όμως χρειαζόταν η πλειοψηφία στο Συμβούλιο Παροδικά ε, γινόταν με ειδική πλειοψηφία αναθεώρηση, όμως από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο και σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά, θα ήθελα να ασχοληθώ με τα μέσα ευελιξίας ε, που μπορούν να κινητοποιηθούν στα πλαίσια του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είπα, για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Υπό την στενή ανέα, όταν εξετάζει κανείς ε, ε, τα μέσα ευελιξία συνειδητοποιεί ότι ε, ο στόχο έχουν να δώσουν μια απάντηση στα χαμηλά περιθώρια που έχουν οριστεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, είναι τα χαμηλότερα από ε, την πρώτη φορά που θεσπίστηκε ε, ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στενά περιθώρια φαινός και η επιθυμία των σύνομοθετών να προγραμματίσουν εκ των προτέρων, εξ αρχής αυτά τα όρια. Οπότε έχουμε περίπου 1% των ορίων για το 2014 έως 2020 που δεν προγραμματίζονται ε, εκ των προτέρων. Ε, κατά 99% προγραμματίζονται εκ των προτέρων όλα τα περιθώρια. Ε, φυσικά υπάρχουν απρόβλεπτες περιστάσεις, δεν χρειάζεται με αυτά που ζούμε να το αναφέρω καν, εξυπακούεται. Επίσης ενδέχεται να αλλάξουν και οι πολιτικές προτεραιότητες διότι η επταετής ε, αυτή περίοδος ε, δεν συμπίπτει με τη θητεία του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως άλλαξαν ε, και άρα αυτοί που προγραμμάτισαν δεν είναι οι ίδιοι που ε, καλούνται να εκτελέσουν το πολιτές σε δημοσιονομικό πλαίσιο εξού και η ανάγκη για τα μέσα ευελιξίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μέσων ευελιξίας ε, στο πολιετές. Τα ειδικά, τα υπονομαζόμενα ειδικά μέσα ευελιξίας καταρχάς, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι ε, στην ετήσια διαδικασία προπολογισμού επιτρέπουν να υπερβούμε τα ανώτατα ωραία. Μπορούν να ψηφιστούν δηλαδή επιπρόσθετα ποσά τόσο στις ε, δεσμεύσεις, ε, στον το, αλλά και στις πιστώσεις πληρωμών. Αυτό πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να γίνεται. Οι πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια γιατί υπάρχει νομική πτυχή και ένας ομιλητής μετά από μένα θα σχολιάσει αυτό το ζήτημα από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να υπερβούμε τα όρια και για τις πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων και τι πιστώσει πληρωμών. Υπήρχαν και στο προηγούμενο πολιετέ αυτά τα μέσα ευελιξία έχουν βαθμονομηθεί, έχουν προσαρμοστεί ε, εκ νέου, όπως βλέπετε τις δύο στήλες, ε, τις έχουν προσαρμόσει στη μέσα μετά το 2013 και το περιθώριο ε, έχει προβλεθεί για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ε, για τις χώρες όπου υπάρχουν κρίσεις ε, ε, σε ονομαστικούς όρους ε, έχει μειωθεί το ποσό για τη βοήθεια αλληλεγγύης αλλά ουσιαστικά είναι υψηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα ποσά είναι για τις φυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κατά ένα χρόνο πλέον το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε ονομαστικούς όρους μειώθηκε όμως παρόλα αυτά είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενη χρήση του για, την, για τις σημαντικές απώλειες είναι αυτό, λόγω της παγκοσμιοποίηση και τρίτον, αλλά και πιο σημαντικό μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού είναι το μέσο ευελιξίας, το flex, το περίφημο, ιδιαίτερα πολύτιμο ε, στοιχείο διότι δεν είναι μετρήσιμο ε, ήδη ε, ετησίω υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια προς το παρόν. Υπάρχει ο σωρευτικός χαρακτήρας και δεν έχει συγκεκριμένο στόχο. Οπότε μπορεί η Δημοσιονομική Αρχή να αποφασίσει πού θα αποδώσει αυτό το κονδύλι και γι' αυτό είναι και τόσο πολύτιμο εργαλείο. Όλα τα μέσα τα έχουμε χρησιμοποιήσει σε ένα ορισμένο βαθμό ε, στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2015 και για το 2016. Βλέπετε τα συγκεκριμένα ποσά στον πίνακα που σας δείχνω. Ε, από ποσοτικής πλευράς ε, η σημαντικότερη χρήση είναι το μέσο ευελιξίας για το 2016, αυτό που ψηφίσατε τώρα πρόσφατα, για τον προϋπολογισμό του 2016 πάνω από 1,5 δις ε, κινητοποιήθηκαν. Έχουμε εξαντλήσει λοιπόν το μέσο για τα πρώτα τρία χρόνια. Στα πλαίσια ε, του τρίτου πακέτου μετανάστευσης, μετανάστευσης migration. Μετά το 2016 θα έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια το χρόνο για το flex και θα αρχίσουμε να ε, ε, έχουμε και πάλι αποθεματικό στα πλαίσια του flex, αλλά προς το παρόν το έχουμε εξαντλήσει για το 2016. Αυτά τα μέσα υπήρχαν όπως ε, έλεγα και προηγουμένως και μας επιτρέπουν να υπεψηφίζουμε επιπρόσθετα ποσά πέραν των ανωτάτων ορίων η εργαλειοθήκη με αυτά τα μέσα ευελιξίας έχει όμως και νέα πολύ σημαντικά μέσα τα οποία παρότι δεν μπορούν, δεν δίνουν τη δυνατότητα αύξησης του συνολικού ποσού, επιτρέπουν παρόλα αυτά την ε, ανακατανομή των πιστώσεων ανάμεσα στα ε, τμήματα και από χρόνο σε χρόνο. Ε, το συνολικό περιθώριο για την ανάληψη υποχρεώσεων για την ανάπτυξη και για την απασχόληση, κυρίως για την απασχόληση των νέων. Μεταφράζει τις προθέσεις του νομοθέτη για αυτό το μέσο και ουσιαστικά επιτρέπει το εξής. Ε, όσα όρια δεν εξαντληθούν μπορούν να σωρεύονται και να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε διαφορετικά τμήματα του προϋπολογισμού. Το νέο μέσο που έχουμε είναι το, περιθώριο, το εφεδρικό ε, περιθώριο contingency margin, ούτω ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις υποχρεώσεων ε, και πληρωμών μέχρι το 0,3% του εθνικού ε, εγχωρίου προϊόντος, 0,03 συγγνώμη, του ακαθάριστου εθνικού ε, ε, εγχωρίου προϊόντος. Και τώρα φτάνουμε προς το παρόν στα 4,4-4,5 δις. Έτσι μπορούμε όχι να αυξήσουμε τα συνολικά ποσά, διότι πρέπει να υπάρξει αντιστάθμιση σε μεταγενέστερα έτη, αφαιρώντας περιθώρια από άλλα έτη. Ε, πρόκειται για ανακατανομή ε, των κονδυλίων, όχι αύξησή τους. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά μέσα ευελιξίας που έχουν ε, άλλα χαρακτηριστικά στη νομοθετική πράξη, στις νομοθετικές πράξεις για τα πολυετή προγράμματα μπορούμε να έχουμε ε, υπέρβαση ή μείωση των κονδυλίων κατά μέχρι και 10% σε ένα συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα ποσά που προβλέπονται ε, στις νομοθετικές πράξεις για τον πολιετή προγραμματισμό. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει ενίσχυση των προγραμμάτων εάν υπάρχει ένα περιθώριο και επιτρέπει εμπροστοβαρή, ε, εμπροστοβαρή χρηματοδότηση, front-loading, back-loading, ε, χρηματοδότηση με διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με τις επιθυμίες ε, αυτών που προγραμματίζουν. Ε, στη συνέχεια, αντιμετώπιση κρίσεων στο γεωργικό τομέα, 400 εκατομμύρια το χρόνο, από τις άμεσες πληρωμές μπαίνουν σε ένα αποθεματικό σε περίπτωση που προκύψει κάποια κρίση και αν τελικά δεν χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό, ε, τότε επιστρέφεται στους γεωργούς. Επίσης, για να σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα για την ε, πιθανή χρήση των νέων μέσων ε, που έχουμε, το εφεδρικό ε, περιθώριο δηλαδή και το περιθώριο για την ανακατανομή, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό των δύο, ούτως ώστε ε, να γίνει ανακατανομή των κονδυλίων ανάμεσα στα τμήματα και από χρόνο σε χρόνο. Παραδείγματος χάρη το συνολικό περιθώριο στον κανονισμό έχει ε, περιοριστεί μέχρι το 2017 για τις πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Εάν όμως θέλει αρχή να ε, χρησιμοποιήσει τα περιθώρια για τα επόμενα χρόνια μετά το 2017 έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει το εφεδρικό περιθώριο ούτω ώστε να τα μεταγενέστερα όρια να τα φέρει σε προηγούμενα έτη και να τα χρησιμοποιήσει για έκτακτες κρίσεις που ενδεχομένως εκδηλωθούν ε, νωρίτερα. Δεν ε, προσφέρουν όμως επιπρόσθετα πόσα δεν πρόκειται για αύξηση κονδυλίων. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται αντιστάθμιση αν χρησιμοποιηθούν νωρίτερα τα κονδύλια ε, μεταγενέστερα συνολικό περιθώριο για τις επιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε χρησιμοποιήσει 2,4 δις για το ΕΦΣΥ, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό έδειξε αμέσως τη δυνατότητα που μας προσφέρει αυτό το νέο μέσο. τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις πληρωμές. Το εφεδρικό περιθώριο έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τούδε μόνο για τις πληρωμές. Κινητοποιήθηκε το 2014 3,2 δις για επιπρόσθετες πληρωμές για να μειωθεί η καθυστέρηση ε, στις πληρωμές ε, ως προς την πολιτική συνοχής και χρειάστηκε να αποφασιστεί αντιστάθμιση ήδη από τώρα ε, για τα χρόνια 2018 έως 20. Ε, ε, τέλος, το επίσης νέο μέσο μέσα στην εργαλειοθήκη μας, το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές GMP. Αυτό μας επιτρέπει και πάλι να έχουμε στη διάθεσή μας ε, τη διαφορά ανάμεσα στο ανώτατο όριο του περιθωρίου ενός χρόνου και, της, ε, του εκταμιευόμενου ποσού της πληρωμής που γίνεται. Το σχεδιάστηκε το περιθώριο αυτό και παρουσιάστηκε από το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές σε δημοσιονομικό πλαίσιο θα δούμε το πλήρες δυναμικό αυτού του μέσου τα επόμενα χρόνια, διότι σε κάποιο βαθμό είναι μια εγγύηση για το ότι ε, όντω μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες τι πληρωμές που προβλέπονται στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά έχουμε και μία μικρή υποσημείωση με αυτή την επιφύλαξη ότι τα τελευταία τρία χρόνια μπορούμε μόνο από 7 έως 10 εκατομμύρια να ανακατανέμουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το χάσμα ε, στις πληρωμές πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο από αυτό το ποσό των 10 εκατομμύριων δηλαδή. Ε, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τις πληρωμές ε, κατά τη διαστολή με το προηγούμενο πολιετές. Ε, θα θυμάστε ότι πάνω από 15 δις σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων τελικά δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν γιατί ήταν σε, δεν ήταν στα σωστά έτη όπου ήταν χαμηλή η απορρόφηση και η εκτέλεση και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στα επόμενα έτη όπου είχε αυξηθεί πάρα πολύ η καθυστέρηση πληρωμές. Το το Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις, όλες οι πιστώσεις ε, ε, και προς το παρόν το 2015 το ποσό ήταν ε, λίγο πάνω από 100 εκατομμύρια και έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται το μέσο και ε, τα επόμενα όμως έτη του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου μπορούμε να δούμε το πλήρες δυναμικό αυτό του μέσου. Εν κατακλείδη. Στόχος και της Κομισιόν και δικό σας στη συζήτηση θα είναι και καθήκον μας να αναλύσουμε την λειτουργία αυτών των οργάνων, να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των οροφών πληρωμών και υπάρχει και μια ακόμα πτυχή, επιθυμώ να σας υπενθυμίσω, που την επεξεργαζόμαστε εντατικά σε σχετικό πλαίσιο, λίγο διαφορετικό, για τον προϋπολογισμό που στοχεύει σε αποτελέσματα. Εργαζόμαστε λοιπόν σκληρά τώρα για την απλοποίηση. Αυτό τι προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις για την απλοποίηση της κινητοποίησης των ε, μέσων ευελιξίας, διότι ορισμένα εξ αυτών είναι δυσκίνητα. Το εξετάζουμε λοιπόν αυτό προσεκτικά, να έχετε υπόψη βεβαίως ότι ίσως χρειαστεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός, δηλαδή ο δημοσιονομικός κανονισμός. Και η διαδικασία αυτή ασφαλώς δεν είναι εύκολη. Όμως, ο αντιπρόεδρος μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ταγμένος σε αυτή την απλοποίηση. Εξετάζουμε τις διαδικασίες και σχετικές προτάσεις μέσα στα πλαίσια της αναθεωρήσεως. Πάλι κάπως περιθωριακά, έχει όμως επίπτωση στην ευελιξία. Η συζήτηση δηλαδή για την επανεξέταση αναθεώρηση θα θέσει πάλι επιτάπητο στο θέμα της διαρκείας του, των μελλοντικών δημοσιονομικών πλαισίων διότι η προβλεψιμότητα είναι βεβαίως άμεσα σχετιζόμενη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας αναπτύξω το θέμα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Σας παρακαλώ να μας διαβιβάσετε το ταχύτερο δυνατό της προτάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το λόγο θα δώσω τώρα στην κυρία Βαλντέρ που είναι τμήματάχης της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για πληρωμές ε, ειδικών μέσων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα περιοριστώ πράγματι σε πέντε λεπτά. Έχετε όλες και όλοι λάβει την ε, γνωμοδότησή μας, ε, η οποία εγκύπτει στο θέμα και γι' αυτό θα σας την αναπτύξω δύο λίγων. Μία προκαταρκτική παρατήρηση πρώτα. Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της κινητοποίησης των ειδικών μέσων πιστώσεων πληρωμών πέραν των ε, περιθωριών, πέραν της οροφής, δεν βρίσκει σύμφωνα όλα τα θεσμικά όργανα. Και υπήρξε η σπαζοκεφαλιά των, ε, των διαπραγματεύσεων του προηγουμένου έτους που τελικά ε, έληξε με δύο μονομερείς δηλώσεις Κοινοβουλίου Συμβουλίου, οι οποίοι τελικώς τα οποία όργανα συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Ας έρθω τώρα στην ανάλυση και ιδίω για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Άρθρο 3, παράγραφος 2 του ΣΕΦΠΕ και επίσης το εκτιμώντας 5 προβλέπουν ότι τα μέσα αυτά μπορούν να κινητοποιηθούν και πέραν των όριων, ε, πέραν των οροφών δηλαδή, των πιστώσεων υποχρεώσεων. Ωστόσο πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δύο ομάδες των ειδικών αυτών μέσων. Τρία από τα μέσα αυτά προβλέπουν ένα μηχανισμό αντιστάθμισης σε ε, βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν τη συνολική οροφή του CFP. Αυτό ισχύει για το περιθώριο απροβλέπτων καθώς και για, το κεφαλαίο, για εκείνα του κεφαλαίου 14 για τη συνολική οροφή δηλαδή των υποχρεώσεων για την απασχόληση και για τα ειδικά κονδύλια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Όσον αφορά τα τέσσερα υπόλοιπα ειδικά μέσα, δηλαδή αποθεματικό για κατεπήγοντα, αλληλεγγύης και ε, μέσω ευελιξίας, δεν τίθεται θέμα αντιστάθμισης. Άρα, συμπεραίνεται ότι όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτά μπορούν να υπερβούν την ανώτατη οροφή CFP. Πρόκειται για ανάλυση βασισμένη στο κείμενο και ενισχύεται και από την πρόθεση, δηλωμένη πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013 που απελευθέρωσε τις διαπραγματεύσεις για το CFP και που λέει καθαρά ότι τα ειδικά μέσα που συζητούνται εκεί υπολογίζονται σε ό,τι αφορά πιστώσεις υποχρεώσεων και εκτός του, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και ευτυχώς ε, την ε, αντίληψη αυτή ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν προκειμένου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τα τέσσερα ειδικά μέσα κινητοποίηση εκτός του πλαφών του CFP e είναι απολύτως δυνατή για πιστώσεις υποχρώσεων. Και τα μέσα αυτά όντως κινητοποιήθηκαν εκτός της οροφής έως τώρα. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν τώρα για τις πιστώσεις πληρωμών. Εδώ δυστυχώς ο κανονισμός ο ίδιος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί ε, το θέμα αυτό στην αναθεώρηση. Το εκτιμώντας 5 και το άρθρο 3 παραγραφός 2 σε ΕΦΠΕ δεν μιλούν παρά μόνο για υπέρβαση των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε ότι το ίδιο το κείμενο του κανονισμού περιλαμβάνει σε δύο περιπτώσεις διατυπώσεις που δείχνουν καθαρά ότι οι πιστώσεις πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πέραν της οροφής CFP. Αυτό συμβαίνει πρώτον για τις αναπομπές που γίνεται στο 4 παράγραφος 1, αυτό 4 παράγραφος 1, για τον υπολογισμό της οροφής των ιδίων πόρων και η οποία πάλι παραπέμπει στο άρθρο 3 παράγραφος 2, η οποία διάταξη δηλαδή παραπέμπει στο 3 παράγραφος 2 και αυτή η παραπομπή είναι σημαντική διότι σημαίνει ότι η κινητοποίηση των ειδικών μέσων για πιστώσεις υποχρεώσεων συνεπιφέρει και πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών πέραν της οροφής του CFP. Εξάλλου, το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού διατυπώνει ρητά ότι εφόσον υπερβεί κανείς την οροφή μπορεί να υπάρξει αυτό, να γίνει αυτό και για τις πιστώσεις υποχρέωσεων και για τις πιστώσεις πληρωμών. Άρα πρόκειται εδώ για οροφή απροβλέπτων. Είναι λοιπόν σαφές για μας ότι η ίδια δυνατότητα κινητοποίησης των ε, κονδυλίων για ε, πιστώσεις πληρωμών πρέπει να ισχύει και για τα άλλα αυτά ειδικά μέσα τα οποία αναφέρονται στο άθρο τελικώς τρια δύο Έχει κάπω τεχνικό χαρακτήρα η παρέμβασή μου, αλλά έτσι είναι. εκτό αυτού, λάβετε υπόψη και τα επιχειρήματα της ορθής, της χρηστής διαχείριση. Στην βάση, οι πληρωμέ ακολουθούν τι υποχρώσεις. Αρχή η οποία καθιερώνεται και με τον κανονισμό CFP, αλλά και από τι αποφάσει για του ίδιου πόρου το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι πιστώσεις υποχρεώσεων υπερβούν την οροφή, οι πιστώσεις πληρωμών πρέπει και αυτές να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πέραν των οροφών, έτσι ώστε να μπορούν να διεξαχθούν σωστά οι πληρωμές. Ε, ε, σε αντίθετη περίπτωση θα προκαλούνταν μια ε, κατάσταση όπου η συνολική οροφή, βλέπετε άρθρο 5 του κανονισμού, θα καταναλωθεί από την χρήση των ειδικών μέσων ενώ το περιθώριο αυτό του άρθρου 5 έχει ε, δημιουργηθεί ειδικά για να διασφαλίζει ότι η οροφή των πληρωμών 9,8 δισεκατομμύρια σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η οροφή των ε, ε, υποχρεώσεων που βρίσκεται στα 960 δις ευρώ. Υπάρχει και το άρθρο 323 τη ε, συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για τον σεβασμό των υποχρεώσεων που έχουν αναλυφθεί απέναντι σε τρίτους. Είναι σαφής εδώ η πρόθεση του νομοθέτου ε, να ε, διαρρήξει αυτή την, αυτό το πολύ στενό περιθώριο με μια μέγιστη ευελιξία ώστε να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις, τους, υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 323 και αυτή η διάταξη απαιτεί ώστε Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή να επαγρυπνούν για την διαθεσιμότητα των κονδυλίων που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρεί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Αυτά μάλιστα είναι λοιπόν, απογραμμένα με χρυσά γράμματα σε μάρμαρο μέσα στα πλαίσια του πλαίσιου του CFP. Διάκριση λοιπόν ανάμεσα σε ε, πιστώσεις υποχρώσεων και πληρωμών με την έννοια ότι η διάσπαση της οροφής μπορεί να ισχύει μόνο για τις πιστώσεις υποχρώσεων θα οδηγούσε σε παραβίαση της ε, ε, εντολής σεβασμού και συμμόρφωσης των υποχρώσεων απέναντι σε τρίτους. Καταλήγουμε λοιπόν ότι το κείμενο του κανονισμού δεν εμποδίζει χρήση των ειδικών μέσων για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και ότι αυτή η κινητοποίηση των ε, πιστώσεων πληρωμών και πέραν της οροφής ανταποκρίνεται στην αρχή της σωστής εγγραφής στον προϋπολισμό αλλά και στην βούληση του νομοθέτου. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος αλλά δεν έχει μικρόφωνο. Σημείωσα ότι δεν θα ήταν υπερβολικά τολμηρό από πλευράς μας να διευκρινίσουμε τα θέματα αυτά. Είναι ενθαρρυντική η γνωμοδότησή σας. Λοιπόν, δέκα λεπτά για ανταλλαγές απόψεων. Ο κύριος Όλμπριχτ πρώτος. Αυτό το συμπέρασμα στην ουσία λέει ότι απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση γιατί τα νομικά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά μεν αλλά κάποιος ε, μπορεί να χαθεί στη λεπτομέρεια. Η γενικότερη πάντως παρατήρηση που κάνουμε είναι ότι η φύση του προβλήματος έγκυται στην αρχή της διατύπωσής του δηλαδή πώς μπορεί οι πληρωμές να ξεπερνούν τις υποχρεώσεις. Και το περιθώριο, ε, θα έλεγα αυτό το πολύ μικρό που έχουμε, είναι 1%, είναι ελάχιστο, δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε διότι αυτό βρίσκεται ε, στην αρχή πάρα πολλών προβλημάτων. Νομίζω ότι η νομική ανάλυση η οποία πρέπει να ακολουθήσει ε, θα δείξει ότι το πρόβλημα με τις υποχρεώσεις δεν υπάρχει. Αντίθετα το πρόβλημα υπάρχει στις πληρωμές. Ε, το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τις πληρωμές. Και έχουμε ένα παλαιό θέμα εδώ με το Συμβούλιο Υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία για το τι μπορούμε να κάνουμε με τη λογική αυτή του Συμβουλίου η οποία λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στις πληρωμές. Ε, λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει η Επιτροπή στην επεξεργασία αυτού του θέματος. Αυτό θα απλοποιήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Και ένα δεύτερο στοιχείο που έχει σημασία είναι <clears throat> να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και η δεύτερη ερώτηση είναι το πότε. Πότε θα εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη συγκυρία που θα μας οδηγήσει στο να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο έκτακτο μέσο. Έχουμε μια σαφή διευκρίνηση των κριτηρίων Ας πούμε η κρίση των προσφύγων είναι μια τέτοια κρίση ή όχι. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε τους σωστούς ορισμούς και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέτω είναι το νομικό κομμάτι της σχέσης πληρωμών και υποχρεώσεων και το δεύτερο είναι το ερώτημα που μόλις έθεσα η κυρία Τόμα και μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για μια πολύ σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Ήταν πλούσιες οι παρεμβάσεις τους και συγκρατώ την ιδέα μιας καλής εφαρμογής του προϋπολογισμού. Έχουμε ένα πρόβλημα με αυτό το πι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι ένα πλαίσιο και σφιχτό πολύ και πιεσμένο πολύ και χαρακτηρίζεται και από σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ύψος των υποχρεώσεων και το ύψος των πληρωμών. Έχουν περάσει ίσα ίσα δύο χρόνια από την αρχή εκτέλεσης του νέου πιδελταπή και ήδη, ούτε σχεδόν δύο χρόνια, ήδη βρισκόμαστε, εάν δεν κάνω λάθος και εδώ είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω, ε, έχουμε εξαντλήσει τα μέσα αυτά τα ειδικά. Ε, βρισκόμαστε στο μέγιστο βαθμό χρήσης, ίσως όχι για τις πληρωμές, αν κατανόησα σωστά αυτό που είπε η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας. Α, συνεπώς λοιπόν αυτή τη στιγμή ψηφιστεί ο τελευταίος προϋπολογισμός βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες δεσμεύσεις για την Τουρκία Οπότε αυτό σημαίνει ότι εκ νέου θα πρέπει να βουτήξουμε πάλι μέσα στον προϋπολογισμό ότι μας χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία μόνιμη δημοσιονομική αναθεώρηση. Δεν ξέρω πού πάμε. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, ένα από τα ερωτήματα, είναι το τι τελικά περιθώριο παραμένει τι δυνατότητα παραμένει για τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας για να κλείσει το πι θα τα βολεύαμε. Αλλά έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας. Και λαμβάνοντας ε, υπόψη την διαδοχή των πολύ σημαντικών κρίσεων, τι έχουμε μπροστά μας. κύριος Λένα για μια πολύ σύντομη απάντηση. Ευχαριστώ σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών άνω του ορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη νομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι πιστώσεις πληρωμών μπορούν να ξεπεράσουν και αυτές τα ανώτατα όρια όπως ακριβώς και οι υποχρεώσεις. Στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μέχρι τώρα τουλάχιστον οι συνθήκες επέτρεψαν το Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αλλού να συμφωνούν, αλλού να διαφωνούν, αλλά να συμβιώνουν μέσω δύο διαφορετικών αναγνώσεων των ε, εναπομεινάντων περιθωρίων. Η δυνατότητα αυτή θα παραμείνει για το μέλλον εφόσον έχουμε βέβαια επαρκή περιθώρια κάτω από τα όρια και ο καθένας μπορεί να βιώνει τη δική του ερμηνεία. Αν βρεθούμε όμως σε μια διαφορετική κατάσταση όπου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα είναι υποχρεωμένα να το ξεκαθαρίσουν το θέμα, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν παράλογο να πρετείνει κανείς μια καλύτερη διευκρίνηση της νομικής βάσης, του νομικού κειμένου. Η αλλαγή όμως του νομικού κειμένου της βάσης απαιτεί ομοφωνία και αυτό σαν εμπόδιο είναι ιδιαίτερο υψηλό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε πριν αναλάβουμε την προσπάθεια αυτή. Πάντως υπάρχει εκεί μια δυνατότητα έτσι ώστε να υπάρξει η διευκρίνηση αυτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα πλαίσια της αναθεώρησης για το τι παραμένει πλέον σε επίπεδο ευελιξίας. Η ε, απάντηση σε αριθμητικό επίπεδο δεν είναι εύκολη. Από τη μία εξαρτάται από το σε ποιον βαθμό και με ποιο τρόπο θα κινητοποιηθούν από τις δημοσιονομικές αρχές τα επόμενα χρόνια τα έκτακτα αυτά μέσα. Σας είπα τι διαθεσιμότητες έχουμε το Flex επανεκκινεί το 2017, ε, οπότε υπάρχει ένα πολύ μικρό περιθώριο. Σε σχέση λοιπόν με τα περιθώρια αυτά υπάρχουν κάποια μικρά μεν, αλλά εξαρτάται από το τι θα ψηφίσετε εσείς και στον επόμενο προϋπολογισμό. Ε, γιατί αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μειώσει και τις, ε, τα περιθώρια για τις πληρωμές. Εξαρτάται λοιπόν και από τις αιτήσει δημοσιονομικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να σας δώσω έναν αριθμό ο οποίος θα ήταν ανεξάρτητος των αποφάσεων που θα λάβετε εσείς στο μέλλον. Κοιτάξτε, μπορέσαμε να αντιχρησιμοποιήσουμε αυτό το περισσόριο ευελιξία το 16 γιατί δεν το χρησιμοποιούσαμε τουλάχιστον στο βαθμό που θέλαμε το 15 και το 14 ο κύριος Φερνάντες. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και για το ίδιο το Συμβούλιο. Δεν έχει πραγματικά καμία σημασία να μιλά κανείς για ευελιξία και να λέμε ότι έτσι κι αλλιώς όλα αυτά υπακούν στους δημοσιονομικούς κανόνες και στον προϋπολογισμό. Όταν μιλάμε για αυτά τα μέσα ευελιξίας τονίζουμε ότι είναι εκτός τακτικής δημοσιονομικής διαδικασίας γιατί αλλιώς τι ευελιξία θα ήταν. Το Συμβούλιο κατανοεί, νομίζω, την επιχειρηματολογία και το πνεύμα ε, της δικής μας ερμηνείας. Εμείς απλά ζητάμε από το Συμβούλιο να προχωρήσει στην σωστή ερμηνεία. Είναι μια δέσμευση την οποία έχει αναλάβει. Δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση να πούμε ότι αποδεχόμεθα ή υποχρεώσεις να είναι μέσα στο προϋπολογισμό και να μην είναι οι συνέπειες, οι πληρωμές. Δηλαδή αυτό ε, δεν έχει πραγματικά λογική. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε το Συμβούλιο να λειτουργήσει με πιο συνεκτικό τρόπο. Μπορούμε να συνδράμουμε ως προς αυτό, μην γελάτε. Και φυσικά τίθεται και το θέμα της γνωμοδότησης της νομικής, ε, την οποία θα κατανοήσει το Συμβούλιο, γιατί γνωρίζει ότι υιοθέτησε 980.000 υποχρεώσεων και 908 ε, ε, πληρωμές. Γι' αυτό ακριβώς οι πληρωμές θα πρέπει να είναι εκτός προϋπολογισμού. Γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση η διαφορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και δεν θα βολεύει κανένα. Και μάλιστα θυμίζω εδώ λέει ο πρόεδρος ότι στο τέλος του 2013 μας περίσευαν προς 203 δις, 203 δις. Οπότε υπάρχουν κάποιοι νέοι παραγόντες κάθε, φορά, κάθε χρόνο τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Όλμπριχτ. Η αίσθησή μου πολιτικά μιλώντας, κατάλαβα αυτά που είπατε και ο, κύριος ε, Φερνάντες τα ξέρει αυτά καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφωνία ε, σε σχέση ε, με τα δημοσιονομικά, διαφωνία ή συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τι σημαίνει όμως διαφωνία και συμφωνία. Υπάρχει διαφωνία ή υπάρχει συμφωνία στις λεπτομέρειες των πληρωμών. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο. Νομίζω ότι στην ουσία είναι σαν να κάνουμε κάτι, να προετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό ελπίζοντας να μην είναι λειτουργικός, να μην πάει καλά. Αυτό είναι μια εντελώς αρνητική αν θέλετε αντίληψη. Αν έχουμε πολύ χαμηλότερες πληρωμές από την αρχή ε, νομίζω ότι το πράγμα δεν θα λειτουργήσει και σε αυτή την περίπτωση θα δικαιωθούμε. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα λίγο πολιτικό σχόλιο. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε τη νομική βάση για να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε, εφόσον βέβαια οι εταίροι βάλουν τα χρήματα. Και μιας και τα χρήματα προέρχονται από τα κράτη-μέλη, πάρα πολύ ε, σύντομα έχουμε ένα θέμα, δημιουργείται ένα θέμα. Πάντως έχουμε χρόνο για να προετοιμαστούμε για το θέμα των πληρωμών. Μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει εύκολα. Περάσαμε από έναν εκ νέου συμπληρωματικό τριγωνικό διάλογο για να το πετύχουμε αυτό. Το επόμενο θέμα το front loading. Προβλέπετε στο άρθρο 15 του κανονισμού για το πολιετές ε, κόσμο, εγγύηση για την νεολαία, ορίζοντας 2020 και ούτω καθεξής. Ε, εκπροσωπούνται ε, δύο γενικές διευθύνσεις, παρακαλώ 8 λεπτά έκαστος, όχι παραπάνω. Ε, νομίζω έχει, έχετε ήδη προετοιμαστεί και ε, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα είσαστε συνοπτικοί. Ο κύριος Κριστόφ που για τον ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Για τον ορίζοντα 2020 θα θυμάστε ότι κατά τη συζήτηση για το πολιετές είχε αποφασιστεί ότι θα εκταμιεύονταν το 2014 200 εκατομμύρια, νωρίτερα δηλαδή, πήραμε από τον προϋπολογισμό 2018, 19 και 20 και τα μεταφέραμε στο 2014. Όπως είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Λένερ, μπορέσαμε να αντισταθμίσουμε τη μείωση ε, και τη διαφορά ανάμεσα στα δύο πολιέτη μέχρι το 2014 και από το 2014 μέχρι το 20. 50% των επιπρόσθετων ποσών, τα 200 εκατομμύρια, τα δώσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Έρευνα και μετά ε, τα υπόλοιπα για τι δραστηριότητα τις δραστηριότητες ε, Marie Λήφθηκε η απόφαση αρκετά αργά το 2014 και ταυτόχρονα εμείς προετοιμάζαμε τον προϋπολογισμό το 2014 και μπορέσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες των δύο ετών αυτών. Ταυτόχρονα υπήρχε και μεγάλη ζήτηση για τα προγράμματα. Το 2013 σας θυμίζω ε, με το backloading ε, είχε το μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με το 2013. 70 ήταν τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν για την έρευνα και για τη Μαρή Κυρή μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις που δεν θα είχαν γίνει διαφορετικά. Κινητικότητα ε, στη βιομηχανία και ε, στα πανεπιστήμια. Τώρα εγκαίρως μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό για το 2015. Τι κάναμε δηλαδή το 2014 και το 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν περίπου 19 δις ευρώ, 13,9 στην βασική μας δράση, πρόταση υποβολής προσφορών και τα άλλα 5,2 δις χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουμε άλλες δράσεις, ΣΔΙΤ, τις ε, κοινέ επιχειρήσεις, άρθρο 185, και τα χρηματοδοτικά μέσα. Α, ναι, και τις διοικητικές δαπάνες. Για την πραγματική ουσιαστική υλοποίηση μετά από δύο χρόνια και μετά από 158 προτάσεις ε, υποβολής προσφορών έχουμε πάρει πάνω από 45.000 επιλέξιμες προτάσεις που ζητούν ε, κονδύλια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρηματοδοτήσαμε πάνω από 6.500 προγράμματα, οπότε 13% ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή μία στις 7 προτάσεις τελικά χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Εάν δούμε τις θετικές αξιολογίες από πλευρά των εμπειρογνωμόνων, φτάνουμε ε, στην αναλογία 1 προς 3. Μία ε, από τις τρεις προτάσεις κρίνουν οι αμερόληπτοι πραγματογνώμονες ότι είναι επιλέξιμη και αξίζει να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ισχυρή ζήτηση στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να εκτελέσουμε το 100% του προϋπολογισμού, είτε πρόκειται για πιστώσεις ανάληψης χρέων, είτε για τις πιστώσεις πληρωμών. Και είμαστε και σχετικά αισιόδοξοι για το τέλος του 2015. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε τον προϋπολογισμό. Ε, τώρα, μόλις ψηφίστηκε ο προπολογισμό το 2016 και κάνουμε τις προβλέψεις μας μέχρι το 2020. Φυσικά γίνονται και οι συζητήσεις για το 2017. Τι προβλέπουμε για τον προϋπολογισμό συνολικό κονδύλι για τον το 2020 περίπου 20,5 δισεκατομμύρια. Τα 14 θα τα χρησιμοποιήσουμε για τις προτάσεις υποβολής προσφορών και τα 6,5 για τις ΣΔΙΤ ε, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού ε, τομέα, ε, διοικητικές δαπάνες Ε, θα πάρετε και τα αποτελέσματα της εξπόστα αξιολόγησης ε, του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα τον Ιανουάριο από ό,τι έχουμε μάθει. Θα έχουμε τα πορίσματα και έτσι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος επί των προτεραιοτήτων που έχουμε για τις σχέσεις με τους πολίτες, για τα προγράμματα δηλαδή. Για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ορίζοντα 2020 προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί πριν ε, το τέλος του 2017. Δεν συμπίπτει με την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, του Πουδουπού. Ναι, ευχαριστώ. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε που ήσασταν και ε, σαφής και συνοπτικός. 5 λεπτά και 29 μιλήσατε. Η κυρία Κριστίνη Στρεμπέρ τώρα για το κόσμο. 8 λεπτά. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Um, very... Με συγχωρείτε, πάτησα το λάθος κουμπί. Σύντομα, για τη γενική εκτέλεση, το 2004 είχαμε φτάσει στο 100% για το financial instrument και σχεδόν 100% για τα υπόλοιπα. Για το 2015 είμαστε πεπισμένες ότι θα τα καταφέρουμε να απορροφήσουμε το 100% μέχρι τέλους του έτους. Εκτός από τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουμε και άλλα σημεία του προγράμματος, έχουμε και ε, προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έχουμε λάβει αιτήσει και γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, αναπτύξω τα δύο πιο σημαντικά, το δίκτυο για τις επιχειρήσεις και το δίκτυο για τους νέους επιχειρηματίες. Εδώ έχουμε προγράμματα COSME δηλαδή και προβλέπεται και εκεί η ενδιάμεση αναθεώρηση 2017. Πρώτη ε, διαφάνεια, Enterprise Europe Network. Αρχίσαμε εκεί από την αρχή του Ιανουαρίου 2015 για 7 χρόνια. Έχουμε ένα αριθμό προτάσεων και χρησιμοποιούμε συμφωνίες πλαίσια για τη συνεργασία και για τη χορήγηση δανείων. Μέσα στο 2014 έχουμε 94 κοινοπραξίες που επιλέξαμε με 559 οργανώσεις, καλύπτουν και τις, ε, ε, τις 28 περιφέρειες και 6 συνεργαζόμενες ε, επιχειρήσεις όπως Αλβανία, Φάιρομ και Άισλαντ. Ισλανδία δηλαδή. Για το 2015-16, εδώ η συμμετοχή της ε, Ένωσης είναι της τάξης του 60%, το ανώτατο όριο δηλαδή. Έχουμε συνολικά ένα ποσό για το 2014-2015 των 100 εκατομμυρίων που θα έχει διατεθεί μέχρι τέλος του 2015 κατά 100%. Η πρώτη ε, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί. Έχει υπογραφεί ένας αριθμός ε, συμβάσεων και για τη δεύτερη έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Έχουμε επιλέξει 12 κοινοπραξίες και προχωρεί η διαδικασία υπογραφών. Μας μένουν τέσσερις προτάσεις, διότι οι ενδιαφερόμενες χώρες, Αρμενία και Ουκρανία, δεν έχουν ακόμα υπογράψει τη Συμφωνία Κόσμη και εμείς αναμένουμε και την κύρωση. Έχουμε και τις πρώτες ε, αξιολογήσεις για τα πρώτες, πρώτους έξι μήνες και δείχνουν ότι καλά τα πάμε. Τώρα ερχόμαστε στο έρασμος για ε, νέους επιχειρηματίες σε αιτήσια βάση και για 24 μήνες. Συνολικά νομίζω είναι σημαντικό να πούμε και να το γνωρίζει το κοινοβόλιο ότι έχουμε πολλά καλά project που μπορούμε ε, που δεν μπορούμε δυστυχώ να χρηματοδοτήσουμε λόγω έλλειψη χρηματοδότησης. Για το 2014 που είμαστε στον 7ο κύκλο μα δηλαδή έχουμε 15 ε, επιλεγμένα project και από τις 28 χώρες που συμμετέχουν στο κόσμο έχουμε 40 project για 14 περίπου εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού. Για το 2015 έχουν επιλεγεί 17 ε, ε, project, σχέδια, με συμμετοχή από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, προϋπολογισμό μας, ήμασταν 5,5 εκατομμύρια για το 2014, είμαστε 7,8 εκατομμύρια το 2015 και χρησιμοποιούμε και την ευελιξία μέσα στο πρόγραμμα COSME και ελπίζουμε ότι θα λάβουμε 8,7 εκατομμύρια για το 2016. Να έρθω τώρα στο χρηματοπιστωτικό μέσο. 60% του συνολικού μας προϋπολογισμού αφιερώνεται στα δύο financial instruments, δηλαδή την εγγύηση δανείων και την equity facility για την ανάπτυξη. Έχουμε χρησιμοποιήσει για το 2014 ολόκληρο τον προϋπολογισμό μας και για υποχρεώσεις και για πληρωμές. Για το 2015 η κατάσταση είναι παρόμοια. Από την πλευρά των υποχρεώσεων 175 εκατομμύρια που αυξάνονται και με συνεισφορές από χώρες ΕΖΕΣ και άλλες που συμμετέχουν και θα ενισχυθούν και άλλο πριν από το τέλος του έτους με πρόσθετο περιθώριο 8,8 εκατομμυρίων από μια μεταφορά η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε από την αρχή του προϋπολογισμού. Και ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή σας Προϋπολογισμών που ενέκρινε τη σχετική μεταφορά πιστώσεως υπέρ του Financial Instrument του κόσμου. Τώρα, από τα εμπροστογεμή ε, front-loading δηλαδή, έχουμε 14 εκατομμύρια για την εγγύηση δανείων υπό την ισχύ του κόσμου. Θα ε, έχουμε ένα πρόσθετο ε, φάκελο 800 εκατομμυρίων που θα, από το οποίο θα ωφεληθούν 12.000 επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του μέσου εγγύησης ε, δανείων. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ω αποτέλεσμα για το 2016 ο διατηθέμενος προϋπολογισμός όπως και για το 2015 δεν θα αποδειχθεί επαρκής για να ε, χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα δάνεια. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου έχουμε υπογράψει 24 συμφωνίες ε, εγγύησης δανείων με 14 χώρες για 263 εκατομμύρια ευρώ. Και υπό, τις, υπό την ισχύ των συμφωνιών έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια που αναμένουμε ότι θα διατεθούν συνολικά υπέρ 180.000 ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια. Και έχουμε και μια πολύ ισχυρή pipeline και τουλάχιστον το 2016 με 30 τουλάχιστον ε, αιτήσει που έχουν ήδη ε, ληφθεί. Ο προπολογισμό καλύπτεται για τα 2015-2017 από εγγύησει που δίνει η ΕΦΣΥ ως μέσα στα πλαίσια του ε, σχεδίου ε, επενδύσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα εγγυήσεων ΕΦΣΥ θα μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες όταν θα έχουμε τον νέο προϋπολογισμό του κόσμου αργότερα. Και για τα έτη 2018 έως 2020, εκεί τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για την αντιστάθμιση του front-loading. Πολύ σύντομα τώρα για την εφαρμογή της Equity Facility for Growth. Βλέπετε την επόμενη διαφάνεια τώρα. Εδώ επισημαίνω ότι σε σύγκριση με το άλλο πρόγραμμα εγγύησης δανείων, εδώ είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση και χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο πριν να μπουν οι πρώτες υπογραφές σε συμφωνίες λόγω του γεγονότος ότι περιλαμβάνονται εκεί και οι ιδιώτες επενδυτές. Η EF πάντως είναι EIF, είναι πολύ δραστηρία και από τον Νοέμβριο του 2015 έχουμε παραπάνω από 7 operations που έχουν λάβει την έγκριση για 86 εκατομμύρια. Πάλι εδώ τα όσα βρίσκονται στον αγωγό, pipeline δηλαδή, προβλέπουν άλλες 6 συναλλαγές για συνολικά 90 εκατομμύρια. Εν ώψη των δεδομένων αυτών, η εφαρμογή της διευκόλυνσης αυτής θα φτάσει στην ταχύτητα που αναμένεται πολύ σύντομα, αρχές του 2016. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο ομιλητή για το Erasmus Plus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για το Erasmus Plus, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο βασίζεται αν θέλετε και αναπτύσσεται στην παλιά πετυχημένη του ιστορία είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεότητα και τον αθλητισμό και περιλαμβάνει απλοποιήσεις ε, σε σχέση με το ενιαίο κόστος και το καεφάπαξα ποσό κόστους. Εφτά διαφορετικά προγράμματα υπήρχαν στο παρελθόν και τώρα περιλαμβάνεται για πρώτη φορά και ο αθλητισμός. Το Erasmus Plus συνεισφέρει άμεσα και στην πρωτοβουλία για τους νέους και την κινητικότητα. Το 70% του προϋπολογισμού αφορά την, την κινητικότητα, προγράμματα που καταπολεμούν την εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης, ε, τον εθελοντισμό και γενικά και την κινητικότητα των νέων εργαζομένων. Εδώ βλέπετε το σχετικό βάρος, το δημοσιονομικό, όπως προβλέψε, προβλέπετε συγγνώμη, στο άρθρο 18 του προϋπολογισμού. Μιλώντας τώρα για το πρότυπο διαχείρισης των ταμείων μας, εμείς χρησιμοποιούμε διαφορετικά χαρακτηριστικά, υβριδικά χαρακτηριστικά. Αλλά έχουμε όμως δύο βασικά χαρακτηριστικά. Έμεση διαχείριση μέσω εθνικών υπηρεσιών και αυτό αφορά το 75% ένας υβριδικός χαρακτήρας sui generis, συνεργασία με τοπικές ομάδες στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας είναι δραστήριο τοπικά και έτσι όμως διασφαλίζουμε μια επικουρικότητα, την, τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και τη συνεκτικότητα του προγράμματος που επηρεάζουν την ευελιξία του. Ο δεύτερος τρόπος διαχείρισης είναι η άμεση διαχείριση μέσω εγκεκριμένων πιστοποιημένων σωμάτων όπως η ΕΑΣΕΑ ή το EIF. 19% ε, το πρώτο και 3,5% το δεύτερο. Και τέλος το μικρότερο κομμάτι είναι άμεση διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα την DG ΕΑΚ και την DG Απασχόληση. Τώρα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έχουμε ένα εξαιρετικό ποσοστό, όπως βλέπετε στους πίνακες, έχετε τους αριθμούς. Παρά προβλήματα εκκίνησης αν θέλετε, καλύψαμε την καθυστέρηση έχουμε ένα ποσοστό σε επίπεδο πληρωμών 100%. θα ξεπεράσουμε το 1,08 δις στις πληρωμές και το 1,07 στις υποχρεώσεις. Το αντίστροφο μάλλον. Καλύτερα από ό,τι πήγαμε το 14. Τώρα για τις πιστώσεις ε, υποχρεω... πληρωμών συγγνώμη, ήταν ένα θέμα που μας ανησύχησε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε κάποια θέματα σε σχέση με την ολοκλήρωση των παλαιότερων προγραμμάτων. Χρειάστηκα το Δεκέμβριο άλλα 108 εκατομμύρια, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ορθή διαχείριση, υγιής διαχείριση. Το 2015 ήταν επίσης δύσκολη λόγω ακριβώς της σορευμένης καθυστέρησης της πληρωμές. Ε, πήραμε άλλα 170 εκατομμύρια τα οποία εκτελούμε στην παρούσα φάση αλλά έχουμε πάει καλά. Ελπίζουμε ότι το 2016 θα έχουμε μία επιστροφή στην κανοτικότητα πρώτη φορά που οι πιστώσεις, ε, ε, τα PA όπως λέμε θα είναι περισσότερα από τα CA, οι πληρωμές περισσότερες από τις υποχρεώσεις. Για το front loading νομίζω ότι είναι κάτι που εφαρμόσαμε σωστά, απορροφήθηκε πλήρως για συγκεκριμένες πολιτικές, ιδιαίτερα όμως για τις δραστηριότητες κατάρτισης και μαθητείας επίσης ε, ένα τρίτο για την ανώτατη εκπαίδευση. The program enables us to uh, biggest impact of the actions we got already in 2014. Υπήρξαν 8.000 προτάσεις ε, το 2014 18.000 προγράμματα επελέγησαν, 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες, 70.000 οργανώσεις και μία μέση διάρκεια των προγραμμάτων από 18, με 2, 18 μήνες βέβαια με 2 χρόνια. Τώρα για το Erasmus Plus λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσδίδει προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχει πολύ θετική επίπτωση στην απασχολησιμότητα και στην κινητικότητα. Ε, Αυξήθηκαν τα εκτήματα απασχολησιμότητας ε, απέναντι στους μη κινητικούς κατά 45%. Ε, η ανεργία για τους φοιτητές του Εράσμους κατά μέσο όρο είναι 23% χαμηλότερη από αυτούς που δεν το χρησιμοποίησαν ε, ήδη έχουμε φτάσει 3 ε, εκατομμύρια κόσμο σε αιτήσια βάση το 16, θα φτάσουμε σε 4 το 20 ε, και τότε ελπίζουμε να φτάσουμε σε 125.000 θεσμικές οργανώσεις. Η υψηλότερη ζήτηση, ψηλότερη υψηλότερη αποφυτικότητα τέλος θα ήθελα να σας μιλήσω για το profiling γενικά <laughs> του προϋπολογισμού μας. Είχαμε κάποιες δυσκολίες ε, στην αρχή του προγράμματος. Υπήρξε μια κάποια απογοήτευση επίσης και δυσφορία. Πήραμε πάρα πολλές αιτήσει τις οποίες δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε αλλά νομίζω ότι για το 2016 η κατάσταση ε, θα είναι ε, πολύ καλύτερη και θα κλείσουμε την περίοδο αυτή με επιτυχία όπως ακριβώς πετύχαμε αντίστοιχες καταστάσεις και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι το Εράσμους, λέει ο Πρόεδρος, είναι ε, μία από τις ναυαρχίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, κάποιον ξέχασα. Η κυρία Σούκοβα Τόιτσεβα για την πρωτοβουλία για τους νέους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πρωτοβουλία για τους νέους είναι 6,5 εκατομμύρια και είναι για την ε, ανεργία των... Ε, ναι, ε συγγνώμη, 6,4 δις ε, και είναι για το ποσοστό ανεργία, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που ξεπερνά και το 25% σε ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει, έχουν προβλεφθεί 34 επιχειρησιακά προγράμματα για 24 επιλέξιμες χώρες. Ε, για το 2014 και για το 2015 τα κονδύλια ε, εκταμιεύθηκαν ε, νωρίτερα με front loading και από τα 6,4 δις χρησιμοποιήσαμε τα περισσότερα τα πρώτα δύο χρόνια. Το 2014 100% εκτέλεση του προϋπολογισμού βάσει των πιστώσεων και το 2015 φτάσαμε μέχρι τον Νοέμβρη 96,23% εκτέλεση. Και ε, η προχρηματοδότηση έχει αυξηθεί για το 2015 και φτάσαμε το 1 δις ε, για το 2014 2020 20 που έχει καταβληθεί στα κράτη-μέλη ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση της πρωτοβουλίας και το 2015 883 ε, εκατομμύρια πληρώθηκαν από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Ενδιάμεσες πληρωμές που έχουμε λάβει μέχρι στιγμή είναι περιορισμένες ε, διότι είναι μεικτή η διαχείριση, με τόσο τρόπος διαχείρισης ε, και η προϋπόθεση να υπάρχει και διορισμένη εθνική αρχή στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαίσιου, πλαισίου ελέγχου. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση, οπότε όταν ε, εγκρίνεται το σύστημα ελέγχου, μπορεί την επόμενη μέρα να ασταλεί η πληρωμή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία καθυστέρηση, στέλνει το κράτος μόνο στην αίτηση και αμέσως γίνεται η πληρωμή. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα Ε, ε, δεν έχουν ορίσει τις αρμόδιες αρχές όλα τα κράτη-μέλη. Η, Ουγγαρία ε, είναι η μόνη που το έχει κάνει, αλλά για τα 29 επιχειρησιακά προγράμματα, επειδή δεν έχει οριστεί αρχή, δεν έχουμε λάβει και τις αιτήσει. Επίσης, 17 εκατομμύρια έχουμε λάβει έτοιμα από την Πορτογαλία. Έχουμε πληρώσει την πρώτη δόση 23,4 και ε, έχουμε και ένα αίτημα για 44,5 ε, εκατομμύρια και θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες. Ε, η Ελλάδα είπε ότι το Δεκέμβρη θα μας στείλει ένα αίτημα για 18 εκατομμύρια γιατί, διότι διόρισαν τώρα την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα και φυσικά θα κάνουμε την πληρωμή. On the για την ε, υλοποίηση των επιχειρησιακών ε, σχεδίων ε, και είναι σημαντικό αυτό για να δείτε το αποτέλεσμα στον προπολογισμό. Το 2014 τα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι είχαν μακροχρόνια ανέργους 110.000, 70.000 ήταν νέοι, Ε, οι 13.400 ε, συνέχισαν ε, την κατάρτιση. 1,3 δίσε συνολικά έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτές τις δράσεις στα κράτη-μέλη μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Δεν είναι ικανοποιητική η απορρόφηση Μπορώ να σας δώσω δεδομένα που πήραμε από τις δραστηριότητες εποπτείας των επιχειρησιακών προγραμμάτων, παρότι δεν έχουμε πάρει τις αιτήσει για αποζημίωση στην Ιταλία. Στις 19 Νοεμβρίου ε, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και πήραμε πληροφορίες ε, βάσει των οποίων ε, ε, ήδη 81% των επιχειρησιακών προγραμμάτων έχει μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις 758.000 ε, νέοι που δεν ε, καταρτίζονται, δεν δουλεύουν, έχουν εγγραφεί στη δικτυακή πύλη και αυτό σημαίνει ότι το 50% των επιλέξιμων έχουν ήδη λάβει μια υποστήριξη. 538.000 έχουν ε, ένα προφίλ, δηλαδή έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους και έχουμε φτιάξει το προφίλ τους, δηλαδή 71% των εγγεγραμμένων νέων, 100.000 ε, Ήδη ε, συμμετέχουν σε δράσεις της εγγύησης για τους νέους, σημαντική αύξηση δηλαδή σε σχέση με τον Απρίλιο, τελευταία φορά που είχαμε δεδομένα και η πλέον σημαντική υποστήριξη πάει σε πρακτικές ασκήσεις. Επίσης υπάρχει μέσο μικροχρηματοδότησης ε, για, τους, ε, για την ε, στήριξη της αυτοαπασχόλησης στους νέους. Για την Ισπανία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ακόμη. Είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος της πρωτοβουλίας για τους νέους με 943 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι 168.000 νέοι είχαν εγγραφεί στη δικτυακή πύλη μέχρι τον Νοέμβρη και μπορώ να σας πω επίσης ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα στην Ισπανία θα τροποποιηθεί και έχουμε λάβει στις 3 Δεκεμβρίου πρόταση τροποποίηση αυτού του προγράμματος και την εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση στη Γαλλία ε, από τους μεγαλύτερους δικαιούχους ε, από μέσα Οκτωβρίου ξέρουμε ότι 77% του προϋπολογισμού ε, είχε ήδη μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις και ε, για τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα έχει εκτελεστεί κατά 80%. Περιμένουμε ακόμη το διορισμό της Εθνικής Αρχής για τα επιχειρησιακά προγράμματα, για το σύστημα υποπτίας και ελέγχου. Έχουμε 32.000 συμμετέχοντες σε δράσεις της πρωτοβουλίες για την νεολαία και ουσιαστικά Αναμένουμε 21% με ε, συμβάσεις πάνω από 6 μήνες όταν ε, ολοκληρώσουν την άσκηση, 19% για ε, συμβάσεις κάτω από 6 μήνες, 5% σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και 33% ακόμη ψάχνουν δουλειά πήρα και τις πληροφορίες για την εφαρμογή στην Πορτογαλία και θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι έχει προχωρήσει αρκετά η Πορτογαλία. Ο συνολικός στόχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι ε, αφορά 33.000 νέους που δεν έχουν ε, needs που δεν δουλεύουν ούτε κάνουν κάποια κατάρτιση 14.000 προς το παρόν έχουν λάβει υποστήριξη, οι, οι μισές είναι οι γυναίκες. και άτομα με ε, αναπηρία ε, και μετανάστες ε, κατά 33%. Ε, επίσης ε, στην, από τους 43.000 που είναι ο στόχος για την πρωτοβουλία, για την, για την επαγγελματική κατάρταση, προς το παρόν έχουμε έρθει σε επαφή με 27.000. Ιταλία, ε, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, μεγαλύτερη δικαιούχοι. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται λοιπόν η υλοποίηση της πρωτοβουλίας ε, και μέχρι το τέλος του 2015 Περιμένουμε την πρώτη αξιολόγηση που γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους και θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το είδος, το εύρος και την ποιότητα των προγραμμάτων. Η βάση του κανονισμού το Μάιο του 2016 θα γίνει η πρώτη ενδιάμεση έκθεση υλοποίηση. Στο μεταξύ όμω θα παίρνουμε τι πληροφορίε από τι Επιτροπές παρακολούθηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση θα πρέπει να υποβάλει έκθεση τον Οκτώβριο του 2016 σε σχέση με την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τη πρωτοβουλία για του νέου Ευχαριστούμε, λέει ο Περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεσή σα ε, για ε, τη συνδιαλλαγή γιατί δεν έχουμε τι πιστώσει για το 2016 αλλά από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση θα δώσουν συνέχεια στο πρόγραμμα, παρότι ακόμη δεν υπάρχουν πιστός. Δεκάλεπτη ανταλλαγή απόψεων, κυρία Τομά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για όλες τις διευκρινήσεις σας. Είναι μια καλή πρωτοβουλία και θα έλεγα ότι οι διαπιστώσεις σας συγκλίνουν και για το Horizon 2020 και για το Erasmus και για το COSME. Είναι παλαιά σε εισαγωγικά προγράμματα, αντίθετα με το Youth Initiative, με την πρωτοβουλία για τους νέους. Διαπιστώνουμε τα σημεία επιτυχίας ακόμα και ξεπερνώντας τα δημοσιονομικά μας όρια. μπορούμε προς στιγμής να ανταποκριθούμε μόνο για το 1 τρίτο για τα προγράμματα που έχουν επιστοποιηθεί και εγκριθεί και έχουν θεωρηθεί επιλέξιμα. Ε, είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Για το Εράσμους είναι χειρότερα ακόμα τα πράγματα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε αν θέλετε σημειώσει για το μέλλον και τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές τις οποίες ε, θα έχουμε στη διάθεσή μας. Θα έπρεπε να είμαστε λοιπόν ευχαριστημένοι από τη διαπίστωση αυτή, αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δημοσιονομικά είμαστε πολύ πιο χαμηλά για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε και για το Εράσμους δυστυχώς είναι κάτι το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε συστηματικά με καθυστερήσεις επίσης συστηματικές. Ένας φοιτητής καθυστερεί να πάρει τα λεφτά του 4-5 μήνες και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το λέγω γιατί θα έπρεπε να είμαστε θεωρητικά ευτυχείς. Δεν είμαστε όμως. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα για το Horizon ε, ε, θα, σταματήσω ε, μια στιγμή μόνο. Για το Horizon 2020 λοιπόν, αντίθετα με αυτά τα οποία είπε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ποτέ δεν επιθύμησε να επανέλθει στη Συμφωνία για την Χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για την Ανάκαμψη. Αντίθετα, εμείς εκφράσαμε την επιθυμία να υπάρξουν μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικές. Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε όμως είναι ότι στο ε, προϋπολογισμό για το πρόγραμμα 2020 και σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε και εσείς και σε σχέση με την πίεση που εμείς εδώ νιώθουμε ε, βλέπουμε ότι θα χρειαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να δούμε ε, κάπως την δυνατότητα αυτή. Το έχετε σκεφτεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Μία επιπλέον ερώτηση για την πρωτοβουλία των νέων. Κοίταξτε είναι ένα νέο πρόγραμμα οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα και απαιτεί περισσότερο χρόνο. Τα λειτουργικά προγράμματα έχουν επικυρωθεί, δεν έχουν επικυρωθεί οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στις αρχές εποπτείας και ελέγχου Ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά ίσως εδώ να με διαψεύσετε. Διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία εγκατάστασης, αν θέλετε. Οι τελευταίες βίδες τώρα μπαίνουν στον μηχανισμό με τις διαχειριστικές αρχές και με τις αρχές ελέγχου και στην ουσία εμείς σταματάμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων για το 16. Αναφερθήκατε βέβαια σε κάποιες εγγύησεις που δόθηκαν για τη συνέχιση της δραστηριότητας αυτής, αλλά είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην σωστή λειτουργία του προγράμματος αυτού και είναι κάτι το οποίο επίσης θα θέσει ερωτηματικά για την συνέχεια του προγράμματος αυτού γιατί κάθε φορά θα πρέπει να περιμένουμε αξιολογήσεις όπως αυτή του 2016. Για τη σχέση ανάμεσα στο Horizon 2020 ε, και τα ΕΦΣΗ έγιναν κάποιες παρατηρήσεις. Για το κόσμο μάλλον θα μιλήσω. Έχει σημασία να δούμε εδώ τη σχέση του με το ΕΦΣΗ στην ουσία αυτό συνιστά το νέο μέσο ευαισθησίας για το κόσμο. Για το Erasmus Plus υπάρχουν δύο στοιχεία που θέλω να θέσω. Όλα φαίνονται θετικά, αλλά η παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μία σόρευση ε, καθυστερημένων. Πόσα είναι αυτά τα καθυστερημένα που δεν έχετε, στα, ε, ε, δεν έχετε σταθεί ικανοί να πληρώσετε αφορά μόνο το Erasmus Plus ή αφορά και τα λεγόμενα DRM, τα μέτρα μείωσης ελλημάτων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε κάθε πολιτική θα έχουμε από εδώ και πέρα DRM τα οποία θα προκαλούν μειώσεις στην προχρηματοδότηση. Είναι τμήμα της νέας πολιτικής ή είναι τμήμα του Εράσμους. Και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι δημοσιονομικό αλλά είναι σημαντικό πρακτικό. Γιατί δεν έχουν ακόμα οριστεί οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι περίπλοκο αυτό, δεν το χρειάζονται. Ε, αν δεν το χρειάζονται τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον το ίδιο το πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Ίσως ακούγεται λίγο αγαθό αυτό που είπα αλλά πρέπει να τύχει απάντησης. Μάνκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα για την πρωτοβουλία για τους νέους, εν συντομία, να πω πως ε, ότι όταν διαπραγματευόμασταν στον τριμερή διάλογο είχαμε πει ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ακόμη για το 2016. Θα καταφέραμε παρόλα αυτά το Δεκέμβρη να πάρουμε τη δέσμευση από τα κράτη-μέλη ε, και ε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Στη χώρα μου... Ε, όταν σταμάτησε η ροή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. 86% των νέων κατάφεραν ε, να βρουν μια θέση εργασίας και μπορέσαμε να μειώσουμε την ανεργία ε, κατά ένα τρίτο. Εάν δεν είχαμε ασκήσει αυτή την πίεση για το 2016 στον τριμερή διάλογο θα μπορούσε να διακοπεί η πρωτοβουλία ε, για τους νέους. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε σε βάθος το ζήτημα, να λαμβάνουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες, γιατί είναι πάρα πολύ καλά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε, κύριε ήθελα να σας ρωτήσω για τον ορίζοντα 2020 και τον αντίκτυπο στο FC. Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το κόσμο. Ξέρω από το δίκτυο επιχειρήσεων πως υπάρχουν προβλήματα όταν περνάμε από επιδοτήσεις χρηματοδοτικά μέσα η αποδάνειες χρηματοδοτικά μέσα. Η προσθετικότητα των κονδυλίων λοιπόν φαίνεται ότι καλύπτει την κατάσταση ή ότι μας λείπει από το ευσύ, καλύπτεται από την προσθετικότητα. Καλά το καταλαβαίνω. Ε, ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα ζητήσω από έναν από τους τέσσερις ε, διευθυντές να απαντήσουν συντομία σε αυτά τα ερωτήματα. Η κυρία την προσθετικοτητα καλα το καταλαβαινω ευχαριστω Λε προεδρος πρέπει να φύγει. Η κυρία Βέρνα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομες ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις για την πλευρά διαχείρισης του έρασμου Συν και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Στην ε, διαφάνεια υπαριθμών τέσσερα. είπατε για το ενδιάμεσο management στο τοπικό επίπεδο είπατε similar του share management δηλαδή συμμετοχική διαχείριση. Είναι το ίδιο όπως τα διαφορετικά ταμεία, δηλαδή εφαρμόζεται η αρχή της ε, κοινή διαχείρισης με κοινωνικούς εταίρους, με ε, τοπικές αρχές κτλ. Ή είναι άλλη μορφή κοινή διαχείρισης. Και τώρα για την απασχόληση των νέων. Υπάρχει κάποια διάδραση, υπάρχει κάποια διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης το οποίο επίσης ε, υποστηρίζει τους νέους όταν ε, χάνει τη δουλειά τους ε, λόγω των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σας ευχαριστώ κύριος Πού. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για το πρώτο ερώτημα της κυρίας Τωμά Νομίζω ναι, ότι με την παρουσίαση προκύπτει πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα και προσπαθούμε να μην αποθαρρύνουμε με αυτό το ποσοστό επιτυχίες ε, τους ε, υποψηφίους που θέλουν να ζητήσουν ε, κονδύλια. Είναι λίγο πρόορη συζήτηση, δεν μπορώ να είμαι πολύ συγκεκριμένος, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα εξετάσει την πρόταση για την αναθεώρηση του, την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορώ να προδικάσω εγώ το τι θα αποφασιστεί. Για το ΕΦΣΥ, ο κύριο Μοέντας, ο επίτροπός μας, το ξεκαθάρισε ότι όταν εγκρίθηκε η πρόταση ΕΦΣΥ, 3% του ορίζοντα 2020 ε, μεταφέρθηκαν στο ΕΦΣΥ δεν χάθηκαν όμως αυτά τα χρήματα από την έρευνα γιατί ε, θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικά προγράμματα και δεν, έχουν, δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος με τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα 2020. Υπάρχει δηλαδή μια συμπληρωματικότητα και όντως θα πρέπει να είμαστε ε, σε επαγρύπνηση ώστε να φροντίσουμε να εκπροσωπούνται ε, δεόντως τα ερευνητικά προγράμματα στο ΕΦΣΥ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπερδέλ που εκπρο... ε, αντικαθιστά, η κυρία Μπερδέλ που ε, εκπροσωπεί την κυρία Σέβερ. Ήθελα να μιλήσω για την αλληλεπίδραση κόσμου και ευσύ και το front loading που γίνεται και στα δύο. Χάρη στο κόσμε ενθαρρύνουμε τους διαμεσολαβητές να, να λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους για τις startup επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, και τους λέμε ότι άμα κάνετε νέα δάνεια 100 εκατομμύρια και περιμένετε απώλειες σε 16% τότε θα καλύψουμε εμείς το 5% των, ε, της προβλεπόμενης ζημιάς τέτοιου είδους συναλλαγές ε, τους προτείνουμε. Οπότε ε, φτιάχνουν το πακέτο δανείων οι διαμεσολαβητές και περιμένουμε να ε, χάσουμε αυτό το κομμάτι από το κόσμο. Δηλαδή είναι το υψηλότερο προφίλ κινδύνο. Αυτό όμως ε, δεν ε, συνάδει με το ΕΦΣΥ γιατί εκεί υπάρχει αντιστάθμιση και δίνουμε δωρεάν εγγυήσει. Ούτε και στο ΕΦΣΥ περιμένουμε να χάσουμε ένα κομμάτι από τις εγγυήσει που δίνουμε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να βασιστούμε στο FC για να ενισχύσουμε την ικανότητα ανάληψης κινδύνου στο κόσμο παροδικά το κάνουμε, αλλά μετά στα επόμενα έτη όλες οι συναλλαγές που προσωρινά καλύπτονται από την ανάληψη κινδύνου του ΕΦΣΥ θα πρέπει να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του κόσμου. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2020 θα είναι αμυγός ε, κόσμε ε, δραστηριότητες, ε, θα απελευθερώσουμε έτσι τον προϋπολογισμό του ΕΦΣΥ και θα χρησιμοποιήσουμε τότε τα κονδύλια για να καλύψουμε άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ε, πάλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Merci, Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καμπαγιό Μπαρασέντας. Merci beaucoup, monsieur le président. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο Όλμπρεχτ, κοιτάξτε, χρησιμοποιήσαμε το σύνολο του δημοσιονομικού μέσου που είχαμε στη διάθεσή μας αλλά όπως είπα και στη διαφάνεια υπαριθμών 6 υπήρξε και ένα κενό ε, στις πιστώσεις ε, ε, υποχρεώσεων και όπως σας είπα πριν πήραμε με 178 εκατομμύρια αλλά το κενό ήταν 200 εκατομμύρια υπάρχει ένα κενό λοιπόν σορεύονται τα χρέη από τη μία χρονιά στην άλλη. Και η δεύτερη ε, ερώτησή σας για τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος και αυτά προκαλούν σωρεύσεις και καθυστερήσεις. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις πιστώσεις υποχρεώ, πιστώσεις υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, όμως ίσως να υπάρξει ένας διορθωτικός προϋπολογισμός, αλλά έτσι και αλλιώς μειώνουμε τη προχρηματοδότηση, ορίζουμε καλύτερα και αυστηρότερα τις προτεραιότητές μας. Merci, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σούκοβα Τούσεβα για το πρόγραμμα πρωτοβουλίας για τους νέους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης ε, όπως τα διευθυντικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι το 2016, 2017 και 18 τα κράτη ε, θα συνεχίσουν να δαπανούν τα χρήματα που είχαν προβλεφτεί το 2015 σύμφωνα με τον κανόνα νήσιν 3. Εμείς στην ουσία θέλουμε να κάνουμε μία αξιολόγηση και να μελετήσουμε μετά το 2017 το πώς πάει το πρόγραμμα αυτό. Είπατε ότι είναι ένα νέο πρόγραμμα, συνεπώς απαιτείται να δούμε σε ποιο βαθμό πετυχαίνει τους στόχους για τον ορισμό των εθνικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε σε σχέση με όλα τα προγράμματα ε, κοινή διαχείρισης. Από τα 400 υπάρχουν μόνο 30 διορισμένες αρχές σε εθνικό επίπεδο και το ποσοστό που καλύπτουμε εμείς εκτός κρατών μελών είναι ένα σύστημα πληροφορικής το οποίο θα συλλέγει στοιχεία εφαρμογής των προγραμμάτων. Έχουμε δημιουργήσει νέους δείκτες και στόχους κοινού για τα ταμεία αυτά και τα λειτουργικά προγράμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως να δημιουργεί πρόβλημα στα κράτη-μέλη και μέχρι τώρα τουλάχιστον ε, εκεί σωρεύεται η καθώς η πλειοψηφία των λειτουργικών προγραμμάτων θα καθοριστούν στις αρχές του επομένου χρόνου. για την ε, διάδραση αν θέλετε με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Όταν ζητάμε ένα πρόγραμμα αναδιάθρωσης από τα κράτη-μέλη Αυτά εξετάζονται από τα γραφεία, από τα σημεία επαφής που έχουμε και βλέπουμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα προγράμματα. Ε, πρόθεση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης ε, ήταν να στηρίξει τους νέους, αν και βέβαια δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ε, τα χρήματα που δίδει το ένα ταμείο με το άλλο, αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον να μην έχουμε επικαλύψεις. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο κομμάτι, το θέμα των πληρωμών, την ώρα της αλήθειας θα έλεγα. Για να μας κάνει την εισαγωγή θα πάρει το λόγο ο κύριος Σιλβάνο Πρέτσα από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω αυτή την παρουσίαση για να σε ενημερώσω για την εκτέλεση των πληρωμών σε σχέση με την έκθεση πεπραγμένων που κάναμε το Σεπτέμβρη. Για το 2015 θα σας μιλήσω για τις προβλέψεις, για τις εκκρεμίες υποχρεώσεις, τα ράλ, τα περίφημα, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Τη γνωρίζετε τη Ζαργκόν. Ε, που χρησιμοποιείται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών βλέπετε τα στοιχεία ανά ε, δαπάνη, ανατμήμα του πολιετούς και θα προσπαθήσω να ε, σας ε, εξηγήσω το γράφημα αυτό. Έχετε δύο γραμμές ε, σε σχήμα ε, νη ε, με δύο διαφορετικά χρώματα, όχι διαγεκομένη. Η συμπαγής γραμμή είναι η πολιτική συνοχής και η πορτοκαλί είναι η γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτή καθορίζει το επίπεδο των εκκρεμιστών υποχρεώσεων γιατί το 2014. Ξεκινάμε, παρουσιάζεται αύξηση για το 2015 και για το 2016. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του αναπρογραμματισμού τμήματος των υποχρεώσεων που είχαν ε, προβλεφθεί αρχικά για το 2014 στον προϋπολογισμό και με τα νέα προγράμματα αυτές ε, οι υποχρεώσεις ε, μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 και εν μέρη και στο 2016. Ε, δηλαδή τεχνητά μειώνεται το ραλ, το υπόλοιπο προς εκαθάριση για το 2014 και στη συνέχεια αυξάνεται τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι λογική αυτή η εξέλιξη διότι οι πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων καταλογίζονται σε κάθε οικονομικό έτος, αλλά μετά ε, υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση για την εκτέλεση των προγραμμάτων και αυτά που πληρώνονται ε, την πρώτη χρονιά είναι οι προκαταβολές και μετά ε, έχουμε τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές. Τι άλλο βλέπουμε σε αυτό το γράφημα. Για τα άλλα τμήματα έχετε τη διακεκομένη ε, κόκκινη γραμμή, τμήμα 1α, σταθερή αύξηση των, ε, του, του ΡΑΛ για το 2014. Στη συνέχεια όμως μειώνεται η αύξηση και σχεδόν το 2015 και 2016 σταθεροποιείται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό για το 2015 και 2016. Τελικά, η απόφαση για το επίπεδο πληρωμών στον προϋπολογισμό κυρίως για το 2016 συνοδεύει την ισχυρή αύξηση των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων και έτσι το 2016 περιερχόμαστε σε μια πολύ πιο άνετη κατάσταση σε σχέση με αυτά που γνωρίσαμε το 2014 και σε ένα ορισμένο βαθμό το 2015. Το ίδιο ισχύει με περαιτέρω βελτίωση το 2016 για τις εξωτερικές δράσεις και το τμήμα 4. Αυτή είναι η διακεκομένη ε, γραμμή με τις τελίτσες στη μέση αύξηση μέχρι το 2014 και 2015. Όμως το 2016 παρατηρείται πως μειώνεται το ράλε οι εκκρεμίες δηλαδή υποχρεώσεις για το τμήμα 4. Πολύ θετικό αυτό, δεδομένου και των περιστάσεων. Μετά, κάτω-κάτω, έχετε τη συμπαγή μπλε γραμμή είναι το οράλι για την κατηγορία 3. Ελαφρά ανωδική η τάση λόγω της σημαντικής αύξησης σε σχετικούς, ε, σχετικούς όρους για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής χρήσης. Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση που σας είπα και παρατηρείται ελαφρά αύξηση για το 2015-2016. Αυτά που έχουν ε, ε, αποδοθεί στον προϋπολογισμό 2014 και εν μέρη και του 2015 επαρκούν για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Για να περάσουμε την επόμενη διαφάνεια. Τέλη Νοεμβρίου. Ε, μας μένει ένας μήνας τι έχει γίνει με την ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου έχουμε 6,7 δις περισσότερες ε, πληρωμές σε σχέση με τον Νοέμβρη του 2014, δύο μονάδες αύξηση για όλες τις διαθέσιμες ε, πληρωμές. Τι σημαίνει αυτό? πως μένουν 11 δις για το Δεκέμβρη, 8% δηλαδή του συνόλου και ξέρουμε πως το Δεκέμβρη, ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχής και για κάποια άλλα προγράμματα, παρατηρούμε πως ε, υπάρχει συσσόρευση ε, ετήσεων πληρωμής για το Δεκέμβρη. Ε, ως προς ε, τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ε, ήταν φυσιολογική η εξέλιξη. Στο πρώτο τμήμα έχετε τη εκταμείωση πολλών κονδυλίων για το Γεωργικό Ταμείο και μετά κατά τη διάρκεια του 2015 σταδιακή και προοδευτική εκτέλεση βάσει του προγράμματος. τι γίνεται τώρα με τα, ε, το στόχο υπερημερίας ε, για τις καθυστερούμενες πληρωμές ε, και την ε, μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, διότι στην άμεση διαχείριση υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις καταβάλλονται επιπρόσθετα οι τόκοι στους δικαιούχους. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τόκοι που καταβλήθησαν ε, ήταν 2,6 ε, εκατομμύρια, περισσότερα δηλαδή σε σχέση με ε, το 2014. 2,2 ήταν πέρυσι, το Νοέμβρη. Μια μικρή αύξηση. Αυτό δείχνει, μια, δείχνει τις ελλείψεις στις πληρωμές όμως τελικά δεν είναι τόσο ανησυχητική η εικόνα, διότι ε, καταβάλαμε αυτούς τους ε, τόκους ε, σχετικά νωρίς το 2015 λόγω των καθυστερήσεων του 2014. Απλώς έγιναν οι πληρωμές στις αρχές του 2015 και βλέπετε ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός καταβολής των τόκων ε, προς τα τέλη του 2015, παραδείγματος χάρη το Σεπτέμβρη και το Νοέμβρη, ε, από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Νοέμβρη για αυτό το τρίμηνο, φτάσαμε 200.000 ευρώ σε τόκους, ενώ ε, στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν τετραπλάσιο το ποσό. Νομίζω λοιπόν ότι επανερχόμαστε ε, σε μια φυσιολογική κατάσταση ως προς την ε, εκτέλεση των πληρωμών. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο επόμενο θέμα. Το περίφημο backlog, οι καθυστερούμενες πληρωμές, το 1β πολιτική συνοχή ε, για τα παλιά προγράμματα. Εκεί υπήρχε μεγαλύτερη καθυστέρηση. Βλέπετε το γράφημα από τις αρχές του 2015 είναι σταθερή η μείωση των ε, αιτήσεων που ε, δεν ε, πληρώθηκαν και βλέπουμε ως ήθιστε τον τελευταίο μήνα έκρηξη διότι έρχονται πολλά αιτήματα το Δεκέμβρη, το τελευταίο δεκαήμερο του χρόνου τις και θα κλείσουμε το 2015 με ένα επίπεδο καθυστερούμενο πληρωμών που θα φτάνει με τα 17 δις. Είναι υψηλό το ποσό, δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε, αλλά είναι μία πρόοδο σε σχέση με τα 20 δις που είχαμε προβλέψει πέρσι. Και συμφωνήσαμε για το σχέδιο πληρωμών φέτος, θυμάστε ότι είναι η προδιαγεγραμμένη πορεία, ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, δεν είναι να έχουμε τόσες καθυστερούμενες πληρωμές. 24 ε, δις είχαμε προβλέψει το 2014 και η μείωση θα είναι ακόμη ισχυρότερη και θα καταφέρουμε να φτάσουμε τα 17 δις ε, μέχρι το τέλος του 2015. Ποιες είναι οι πρόπτικες για το 2016? Για το 2016 Θεωρούμε ότι αυτή η αδικαιολόγητη ε, καθυστέρηση ως προς πληρωμές για το 2014 και το 2015 ε, τελικά θα εξομαλυνθεί και το 2016 θα έχουμε δύο δις καθυστερούμενων πληρωμών. Είτε διότι ε, οι αιτήσει έρχονται τελευταία στιγμή και δεν μπορούμε να τις διεκπαιρεώσουμε, δεν προλαβαίνουμε, ή υπάρχει μια διακοπή διότι χρειάζεται να ε, διεξαχθεί κάποιος έλεγχος. Για την τήρηση του προγράμματος πληρωμών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λοιπόν. Και για το 2016 με τις ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα μπορέσουμε να καλύψουμε ακόμη και τα έκτακτα μέτρα για την Ελλάδα με front-loading, προκαταβολή των ποσών. Θα καλύψουμε επίσης και τα αιτήματα αποζημίωσης των νέων προγραμμάτων 2014 ε, για τον ορίζοντα 2020. Είναι ήδη συμπεράσματος, θα έλεγα ότι όλο ένα και απομακρυνόμαστε από την κρίση που εκδηλώθηκε το 2014, ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση το 2015 και όπως πηγαίνουν τα πράγματα τώρα, θα επανέλθουμε στη φυσιολογική κατάσταση το 2016 και μπορούμε απρόσκοπτα να ε, προχωρήσουμε με την εκτέλεση των πληρωμών. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέζε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για τις καλές προοπτικές που δώσατε. Κύριε Όλμπριχτ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα για τις, ε, τα, επιτόκια τους στόκους υπερημερίας. Υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρών μελών. Χώρε μέλη και δικαιούχοι από την άλλη μεριά. Δεν τα έχουμε αυτά στη στατιστική ή δεν υπάρχουν. Δεν τα έχουμε στη στατιστική ή δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Δεύτερο. Δεύτερο ερώτημα λέτε ότι προς τα τέλη του 2016 θα έχετε δύο δις. Πώς θα γίνει αυτό και τι γίνεται με το 17 και το 18. Διότι 2 δισεκατομμύρια το 16 θα επανέλθουμε το 17-18 ή θα κρατήσουμε το 2%. Γνωρίζω ότι 2 είναι οι παλές καθυστερήσεις τι γίνεται με τις νέες καθυστερήσεις, backlog δηλαδή. Είναι ενδεχόμενο να υπάρχει αυτό και είπατε ότι φτάνει το 95% του κατοφλίου. Τι γίνεται με το 5% εάν λάβετε δηλαδή και αυτό υπόψη. Κύριε Τωμά. Σας ευχαριστώ. Είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι μειώνονται οι τόκοι ε, για τις καθυστερήσεις. Είναι κάποια παρηγοριά. Για να ρωτήσω όπως και ο κύριος Όλμπριχτ. Αυτή η κάπως αισιόδοξη προοπτική που μας περιγράφεται μήπως προέρχεται από το γεγονός ότι τα 20 δισεκατομμύρια που προβλέπονταν αρχικά το για το 2016 αντί των 17 μήπως είναι κάπως και συνέπεια του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα ήταν πολύ καθυστερημένα και ότι τελικά οι αιτήσει πληρωμών έρχονται και αυτές με καθυστέρηση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Α, δεν βλέπω. Α, εσείς κύριε Μάνκα. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Συντομότατα έχω να ερωτήσω το εξής. Εάν, εφόσον μάλλον, η εφαρμογή έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα, τέλη του 2016, ποιες πληρωμές θα εκκρεμούν ακόμη, δηλαδή ποιες, υποχρε... ποιες ποιοι ε, λογαριασμοί θα εκκρεμούν ακόμη, θα είναι ακόμη απλήρωτοι. Ευχαριστώ εσείς τώρα κύριε Ρεζά. Για να απαντήσετε τις ερωτήσεις ε, των εισηγητών μας και του κύριου Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ερώτηση Όλμπριχτ. Όντως, κατά κάποιο τρόπο, το αποτέλεσμα των τόκων των καθυστερημένων πλωμών εφαρμόζονται μόνο στο direct management, όταν δηλαδή οι δικαιούχοι είναι άμεση αντισυμβαλόμενοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ισχύει όπου η εφαρμογή, η implementation δηλαδή γίνεται μέσα των χωρών μελών. Υπάρχουν δηλαδή οργανισμοί στις χώρες μέλη που τα εφαρμόζουν. Αυτά λέει και ο κανονισμός, αυτοί είναι και οι συμφωνημένοι κανόνες και είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβαστούμε. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε το 2014 και 2015 να διαχειριστεί με ενεργό τρόπο τις διαθεσιμότητες των πληρωμών έτσι ώστε να περιορίσει τις πληρωμές τόκων καθυστερήσεων, διότι δεν είναι τρόπος να δαπανάτε έτσι το σπάνιο δημόσιο χρήμα. και για την κοινή διαχείριση με χώρε μέλη, αν ήταν μόνο κοινή διαχείριση με μέλη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όπως είμαστε τώρα, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, νομίζω ότι για του χρόνου ο στόχος της ελαχιστοποίησης, δηλαδή να μην χρειάζεται να πληθωρωθούν καν τόκοι για καθυστερημένες πληρωμές, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να συμμορφωθεί με όλες τις ε, σημαντικές της υποχρώσεις, είναι εύλογο σενάριο, δηλαδή είναι δυνατόν πράγματι να ελοπιθεί Τώρα, τι γίνεται με τις καθυστερούμενες πληρωμές των 2 δις που αναμένονται για το 2017 και 2018 για τα προγράμματα συνοχής και πέραν το 2016. Αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε σταδιακά να τις καταργήσουμε τελείως μέχρι το 2017. Θα εξαρτηθεί αυτό από το πόσες χώρες μέλη θα φτάσουν στο κατόφλιο του 95% μέχρι τότε. Θα είναι και η διαδικασία κλεισίματος που θα χρειαστεί κάποια προσπάθεια και κάποιο χρόνο. Πάντως η πρόβλεψη για την ώρα είναι ότι θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το εναπομένων 5% στο 2017 ή στα επόμενα χρόνια. Για τις πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις είμαστε σε θέση επί του παρόντος να δούμε πιο καθαρά για το 2016 οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2017 είναι και αυτές μάλλον αισιόδοξε από την άποψη αυτή αλλά για να έχουμε πλήρη εικόνα του δημοσιονομικού πλαισίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει την επόμενη άνοιξη για να μπορεί να λάβει υπόψη και ένα άλλο στοιχείο που είναι η τεχνική προσαρμογή που μένει να γίνει για την πολιτική συνοχή έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην σχετική ανάπτυξη των χωρών μελών, ώστε θα χρειαστεί ορισμένα στοιχεία να προσαρμοστούν. Όταν θα είναι σαφές το στοιχείο αυτό και θα υπάρχουν οι σχετικές στατιστικές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να προσφέρει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση κυρίας Τόμα, είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα λόγω του ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής και αλλού. Η ερώτηση είναι ναι. Ε, η συγγνώμη, απάντηση είναι ναι. Αν είχαμε συνεχίσει με πλήρη ταχύτητα, θα ήμασταν σε πιο δύσκολη κατάσταση για το 2016. Τούτου λεχθέντος πάντως, υπενθυμίζω ότι στον προϋπολογισμό του 2016, όσο έχει τώρα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα περιθώριο των 2 δισεκατομμυρίων στις πληρωμές, σύμφωνα με την κοινή ερμηνεία που δίνει Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και αν είχε γίνει λοιπόν ταχύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων, θα, θα υπήρχε κάποιο περιθώριο. Τώρα, για την ερώτηση Μάνκα, για το επίπεδο των υπολείπων προς εκαθάριση για το τέλος του έτους. Στα τέλη του 2015 το επίπεδο των εκκρεμών υποχρεώσεων θα είναι 217 δισεκατομμύρια. Δύο τρίτα από αυτά πολιτική συνοχής. Στο τέλος του 2016 θα αυξηθεί το ποσό αυτό κατά 11, 11 Κατά 11 δις. Δηλαδή θα πάει στα 228 δις στα τέλη του 2016. Αυτή η αύξηση του 2016 αποτελεί τη διαφορά μεταξύ υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό το 2016 και του συνολικού επίπεδου πληρωμών. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στα δύο, αυτό ποσά, τα δύο αυτά ποσά θα είναι αυτή που θα προσθεθεί. Αυτά βέβαια με την, υπό, υπό την υπόθεση ότι δεν θα προσθεθούν και άλλες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Ζά. Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης αυτής συνάντησης του monitoring στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επειδή ο κ. Όλμπριχτ ε, έκανε την εισαγωγή αρχικά, η κυρία Τωμά ας προβεί στην συναγωγή των συμπερασμάτων. Θα ήταν φιλόδοξο από πλευρά μου να προτείνω ένα συμπέρασμα σε αυτή τη φάση των συζητήσεων. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο για την ειλικρίνειά τους, την ευκρίνειά τους. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα καθησυχασμένη σε σχέση με το PDP. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε λέγοντας ότι ορισμένα πολύ σημαντικά προγράμματα, ιδιαίτερα δημοφιλή, ήταν υποχρηματοδοτούμενα σε σχέση με τις προσδοκίες που υπήρχαν. Δεύτερον θα ήθελα να παρατηρήσω ότι για πρώτη φορά σταματάμε ουσιαστικά ένα πρόγραμμα πριν από την αξιολόγησή του και αναφέρουμε εδώ στην πρωτοβουλία των νέων. Πάντως είναι πρώτη φορά που σταματάμε τις υποχρεώσεις για ένα πρόγραμμα σε σχέση με ε, την αξιολόγησή του. Είναι ένα νέο δυναμικό πρόγραμμα όμως το οποίο αφορά στους νέους και στο μέλλον μας. Τρίτο σημείο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε ήδη, είναι το θέμα των πληρωμών. Πάντα περιμένουμε να γίνει το θαύμα, πάντα περιμένουμε να μην έρχονται πολύ νωρίς οι υποχρεώσεις Υπάρχουν γενικά πολλά προβλήματα τα οποία ε, εξαρτώνται από την τύχη. Η τύχη όμως δεν υπηρετεί πάντα την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στον κλάδο των επενδύσεων, ούτε στον κλάδο της ανάκαμψης, ούτε στο θέμα της ευμάρειας των πολιτών γενικά. Όλα αυτά ουσιαστικά αποτελούν δυσλειτουργίες ε, οι οποίες ορεύονται, δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του νέου πιδελταπή Ευχαριστώ και για τις ε, νομικές διευκρινήσεις που έχουν δοθεί σε σχέση με τα ανώτατα όρια για τις πληρωμές και κατανοώ βέβαια ότι ο κανόνας της ε, ομοφωνίας κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα αλλά πάντως αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και θα πρέπει να παρετηθούμε τότε δεν θα πάμε πουθενά διαπιστώνουμε το βαθμό δυσκολίας αλλά πιστεύοντας στην Ευρώπη και με τον βολονταρισμό που μας χαρακτηρίζει θα μετακινήσουμε ακόμα και βουνά. Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λέει ο πρόεδρος την κυρία Τόμα. Ε, συνάδελφοι, μιας και ήρθατε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Προϋπολογισμών, δεν διαλέξατε τα εύκολα. Οι προϋπολογισμοί είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Ευχαριστώ λοιπόν τους προσκεκλημένους που τόσο μας διαφώτισαν, που μας έδωσαν την δυνατότητα να λειτουργήσουμε κι εμείς με ευκρίνεια, Δεν θα προσπαθήσω να είμαι υπερβολικά τολμηρός και εγώ προσπαθώντας να διευκρινίσουμε την δυνατότητα του να ξεπεράσουμε τα όρια για τα διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα που συζητάμε είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα και σε μια συμφωνία και μιας και οι χώρες μέλη συμμετέχουν στη συμφωνία, τότε θα πρέπει και οι δύο επί του προϋπολογισμού αρχές να συμφωνήσουν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ τους συναδέλφους από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Είμαι σίγουρος ότι ενδιαφερθήκατε για αυτή την σημαντική στιγμή συζήτησης. 27 Ιανουαρίου η επόμενη συνάντηση του Monitoring Group θα αναλύσουμε τον ορίζοντα 2020 και το Connecting Europe. Περνάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν της ημερίστιας διάταξης. Τώρα είναι οι ψηφοφορίες. Je vous invite à glisser vos cartes à dans les appareils de vote. Ετοιμάστε, ετοιμάστε τις κάρτες σας για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μικρό τεστ πριν ξεκινήσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Bien, le scrutin est ouvert.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 Λοιπόν, τρει από εσά ή δεν ψηφίσατε ή τα μηχανάκια σα δεν δουλεύουν. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Νεγκρέσκου για την κινητοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για την Ιρλανδία. Η τροπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη 13 κατά 12 υπέρ. 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη 14 κατά 11 υπέρ. 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5 υπέρ κατά απερίφθη. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται δεκτή 15 υπέρ 8 κατά 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 10 υπέρ κατά δεκτή. 11 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. Δεκτή 13 υπέρ 12 κατά. 12 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. δεκτή 13 υπέρ κατά δεκτή 14 υπέρ κατά δεκτή 15 υπέρ qui est contre Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15 ψηφίζεται. Άρχεται η συνεδρίαση. Τέλος. Δεκτή 12 υπέρ 9 κατά 4 αποχές. 16 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή για το σύνολο του κειμένου τροπολογημένου με ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτό. 18 υπέρ 6 κατά. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τζάνι για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης Φιλανδία. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτή έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή επτά υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 8 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία τέλος δεκτή 9 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή Δέκα υπέρ κατά αποχές δεκτή Εντέκα υπέρ κατά αποχές δεκτή Δώδεκα υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Για το σύνολο του κειμένου τροπολογημένου με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Δεκτή 21 υπέρ, 4 κατά. Περτάμε τώρα στην έκθεση Zabal Rubial για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ετήσια έκθεση. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Α, ζητήθηκε έλεγχος για την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 14 υπέρ 12 κατά. Τώρα τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α για, συγγνώμη, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5. Τέλος. 13 υπέρ, δεκατρεις κατά. Απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Απορρίπτεται 14 υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 7 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας, δεκτό το δεύτερο τμήμα, 15 υπέρ 11 κατά. Τροπολογία 9, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, 10 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Λοιπόν, για την τροπολογία υπαρίθμου 10. Η 9 έγινε δεκτή. Η 10 λοιπόν. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Δεκτή. 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 14 υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 12 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 17. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 14 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επί του συνόλου του κειμένου ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται Τέλος. 20 υπέρ 4 κατά 2 αποχές. Περνάμε λοιπόν τώρα στις μεταφορές στον προϋπολογισμό. Τρίτο τμήμα, προϋπολογισμός 15, η κυρία Ζάβαλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έχουμε πολλαπλές μεταφορές, τη 36 και 39 για την παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που ψηφίσαμε. Και 42, 43, 44 και 45 για την ανθρωπιστική βοήθεια 12 εκατομμύρια για το Αφγανιστάν, 20 εκατομμύρια για το Σουδάν του Νότου, 15 για την Ιεμένη και 13 για τη Σερβία και την Μακεδονία λέει ο Μιλήτρια. Καλώς, ευχαριστώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά για τις τέσσερις αυτές μεταφορές. Δεν έχετε αντίρρηση. Ονομαστική πλήση. Κοιτάξτε, έχουμε καταρχάς τα δύο, τις δύο πρώτες μεταφορές 40, 42 και 45 λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε τις δύο για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και μετά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θα πρέπει να αναμίξουμε τις δύο κατηγορίες. Καλώς λοιπόν η 36 και 39 λέει τώρα ο Πρόεδρος ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Λοιπόν 22 υπέρ 4 κατά. Και τώρα 42 με 45. 42, 43, 44, 45. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 24 υπέρ 2 κατά. Τώρα περνάμε στην κυρία Χολμάιερ για τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω διότι την προηγούμενη φορά μου είχατε να μου είχατε ζητήσει να σας λέω τα νούμερα τώρα μου είπατε να μην σας τα λέω βεβαίως ο καθένας μπορεί και να τα διαβάσει στο έγγραφο αν μου ζητήσετε να σας, το, να σας τα λέω τα νούμερα τότε πάλι θα το κάνω την επόμενη φορά Ε, κάθε φορά κάποιος παραπονείται και για κάτι άλλο. Τώρα, EP Transfer και το σε 6 πρόκειται για τις συνεισφορές για τα ευρωπαϊκά σχολεία. 85.000 από το αποθεματικό για απρόβλεπτα. Κεφάλαιο 27. Δεύτερο, μεταφορά που έχει κάποιο νόημα δηλαδή τα χρήματα που μένουν αδιάθετα στο τέλος του χρόνου να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας που ε, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για του χρόνου επομένως. Αν βλέπω λοιπόν καλά πρόκειται για 71 εκατομμύρια για να ε, αποπληρωθούν πρόωρα ορισμένες ε, υποχρεώσεις έτσι ώστε να μην ε, είναι καταβλητή η τόκη περιμερίας. Αυτό ήταν όλο. Καλή χρήση, λέει ο Πρόεδρος, των ε, χρημάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν πρόκειται για ένα είδους επενδύσεως. Και βλέπετε κιόλας και κατά πόσον το δημοσιονομικό μας πλαίσιο μας καταδικάζει να κάνουμε ορισμένα πράγματα διότι όταν λήφθηκε η απόφαση να γίνει δηλαδή η επένδυση σε αυτό το κτίριο Κόνραντ Αντενάουερ θα έπρεπε να έχει εγγραφεί ως επένδυση στον προϋπολογισμό. Αλλά επειδή έχουμε αυτό το περίφημο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναγκαζόμαστε να κάνουμε τέτοιες διαχειρίσεις που δεν είναι ορθές κατά γράμμα. Έτσι πρέπει να λέμε κάθε φορά ότι εν ώψη των περιορισμών που ε, υφιστάμεθα κτλ. Να πούμε λοιπόν πρώτα για την ε, πρώτη μεταφορά για τα ευρωπαϊκά σχολεία που οφείλεται εν μέρη και στο γεγονός ότι ορισμένοι ε, συνεργάτες έχουν δικαίωμα να ε, στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έχουμε λοιπόν αυτή την υπαριθμό σε 6 με ονομαστική ψηφοφορία και αρχίζει η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ. Λείπει μία ψήφος ακόμη. Τέλος. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Για την δεύτερη μεταφορά, σε 7 2015, για το κτίριο CAD, 71 εκατομμύρια. Αρχίζει η ψηφοφορία, πάλι ονομαστική. Πέρας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Για τα ακίνητα, πολιτική ακινήτων, για το κτίριο της οδού Μόντου Αγία, κυρία Χολμάιερ. Θα προσπαθήσω και εδώ να είμαι σύντομη. Πρόκειται για το εξή. Έχουμε ένα κέντρο εκπαιδεύσεως, το οποίο έως τώρα ήταν εγκατεστημένο στο κτίριο της οδού ΑΓΕ 63. Το κτίριο αυτό έχει άμεση, επίγουσα ανάγκη ανανεώσεως, ανακαινήσεως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αναγκάζεται να βρει κάποια λύση ε, που να είναι βιώσιμη για το μέλλον. Οι ετήσιες δαπάνες για το κτίριο της οδού Μοντουαγέ 63 ανέρχονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια. Συνολικά όλα μαζί. Για το 2016 θα καταβάλουμε το μισό μίστομα, αλλά θα πληρώσουμε το κόστος για όλο τον χρόνο, τα άλλα κόστη δηλαδή, καθώς και για φόρους και για την περαιτέρω συντήρηση, διότι η σύμβαση λίγοι τα τέλη του 2016. Ωστόσο, δείχνει κατανόηση ο ιδιοκτήτης, διότι μας επιτρέπει προσωρινά να μετακομίσουμε σε άλλο κτίριο δικής του ιδιοκτησίας. Και θα πληρώσουμε μόνο το μισό μίσθωμα, 720.000 ευρώ για το άλλο μίσθωμα δηλαδή. Για το 2016 θα πληρώσουμε εκεί και τους μισούς φόρους. Γιατί για το άλλο κτίριο πληρώνουμε ολόκληρους τους φόρους είναι διότι η σύμβαση μισθώσεως λήγει το 2016. Και έχουμε στην κατοχή μας το κτίριο για όλο αυτό το διάστημα. Στο άλλο κτίριο θα έχουμε λοιπόν μειωμένα, μειωμένες δαπάνες. Έχουμε όμως βέβαια δαπάνες της μετακομίσεως της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Χρειάζονται και κάποια έπιπλα για τη μεταβατική περίοδο, 200.000 και χρειαζόμαστε άλλες 400.000 για, άλλα, ε, για, άλλο εξοπλισμό. Καλούμεθα να μετακομίσουμε σε άλλο μεταβατικό κτίριο γιατί αλλιώς δεν θα ήταν δυνατό να γίνει ανακαίνιση του πρώτου κτιρίου ανακαίνιση την οποία αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, θα το κατεδαφίσει το κτίριο και στο μεταβατικό θα παραμείνουμε και το 2017, στη διάρκεια του οποίου θα ανεγερθεί ξανά το πρώτο κτίριο. Γι' αυτό το 2017, μαζί με όλα τα κόστη των 3,2 εκατομμυρίων, από την άποψη τετραγωνικών μέτρων, το κτίριο στο οποίο θα μετακομίσουμε είναι περίπου το ίδιο, τα 3,2 εκατομμύρια αντιστοιχούν περίπου στο ύψος του κόστους του προηγούμενου. Για το 2018 θα χρειαστεί να πληρώσουμε ακόμη το 1 τέταρτο των δαπανών για το μεταβατικό κτίριο. Θα έρθουν βέβαια και οι δαπάνες για τη μετακόμιση τη τάξη των 4,275.000, 4.275.000 και ε, δεν είναι δυνατόν να αποφευθούν. Όμως η διοίκηση του Κοινοβουλίου κατόρθωσε το κόστος για την μίσθωση του κτηρίου, το οποίο θα είναι απολύτως νέο κτηρίο βεβαίως έτσι, να το διατηρήσει στο ίδιο ύψος. Νομίζω ότι τελικά είναι λογική η ρύθμιση. Θα πάμε λοιπόν για το ενδιάμεσο διάστημα στο κτίριο της οδού Μπελμονκούρ και θα επανέλθουμε το 2017 στο κτίριο της οδού Μοντοαγία, το οποίο θα είναι ολοκένουργιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας και οι δαπάνες που θα αντιμετωπίσουμε δεν θα είναι υψηλότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Ε, κάπου κάπου βέβαια πρέπει να ε, ανακαινίζουν τα κτίρια, δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εξήγηση που δώσατε. Έχετε ερωτήσεις μήπως, κάποιος εξημών. Όχι. Άρα, στη βάση της ε, ε, θέμα του θέματος από θα Χολμάιερ, καλούμεθα να λάβουμε θετική απόφαση. Μπορεί να γίνει και διανατάσσεω τη χειρό. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχέ. Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή προεπολισμών τάσεται υπέρ του εγχειρήματο. Έχαμε προβλέψει για τις 11.45 αρχικός παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, αποφάσεως να ε, διαθέσει 3, 3, 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Το λέω αυτό διότι είναι ακριβώς 11.45. Πολύ καλά λοιπόν. Και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ότι όλες και όλοι τηρήσατε τον χρόνο που σας είχε δοθεί. Με μεγάλη υπομονησία αναμένουμε τώρα την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως ο Χωσέ Μανουέλ θα με διορθώσει εάν χρειαστεί. Ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του προϋπολογισμού 2016 έχει εγκριθεί ε, στις 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης ο προϋπολογισμός του το 2016 και στις 29 Νοεμβρίου μάθαμε ότι το Συμβούλιο μετά από πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει να ε, διαθέσει 3 δις στην Τουρκία. Αν εξετάσετε τώρα τον ψηφιστέντα προϋπολογισμό του 2016 δεν θα βρείτε ίχνος των 3 δισεκατομμυρίων. Άρα μας απασχολεί το θέμα. Και όταν λέω ότι ανυπομονούμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέω διότι είδαμε και ε, κάποιες πρωτοβουλίε ε, trans funds καταπιστευμάτων για την Συρία, για την Αφρική. Ε, αυτά είναι δημοσιονομικοί δορυφόροι του προϋπολογισμού που εν μέρη χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και καλούνται εν, ε, κατόπιν και οι χώρες μέλη να συνεισφέρουν και αυτό πρέπει να είναι εξασφαλισμένο και όλες, ε, όλοι αυτοί οι δορυφόροι είναι στην πραγματικότητα ε, παραμορφώσεις του ευρωπαϊκού ε, και τώρα μας προτείνουν τρία για την Σύρια λέει ο ε, αλλά όταν προσπαθήσετε να εξηγήσετε στους συμπολίτες σας τι πάει να πει ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πρέπει να έχετε στέρεα επιχειρήματα για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι άνθρωποι τι τους λέτε. Ή οσδήποτε δημοκρατικός θεσμός πρέπει πρωτίστως ε, να καθιστά τον ε, ε, προϋπολογισμό του διαφανή και στα όματα των, των πολιτών. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που τα εξήγησαν σήμερα οι κύριοι Ολμπρίχτ και Τόμα και μα επιτρέπει αυτό, μα έχει επιτρέψει δηλαδή, η προσπάθεια αυτή να κάνουμε και κάποιε πρόοδου. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στο πρόσωπο τη κύρια Καλβίνιο που είναι η Γενική Διευθύντρια και στην οποία ε, ευχαρίστω ε, παραπολώ το μικρόφωνο. The floor στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλές πληροφορίες και πάντοτε είναι καλό να ερχόμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρξουν ε, παρανοήσεις. Θα τα πω στα αγγλικά. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας ότι η προσφυγική κρίση ήταν ε, η μεγάλη σκιά ε, πάνω από τα κεφάλια μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και δεν ξαφνιάζεται κανένας. Φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε εξάλλου πώς θα ανακύψουν νέες ανάγκες για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την ε, ιστορική σημασία ε, κρίση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό έγινε ήδη μεγάλη προσπάθεια και από πλευρά Κοινοβουλίου και από πλευρά Συμβουλίου και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί επιμείνατε γι' αυτό. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν τα τμήματα του προπολογισμού που είναι στο πρώτο μέτωπο ε, για την αντιμετώπιση τη κρίση. Τμήματα 3 και 4 συγκεκριμένα διπλασιάσαμε του πόρου μπορούμε να κινητοποιήσουμε από 2,4 δις φτάσαμε σχεδόν τα 9 για τα χρόνια 2015 και 2016. Γνωρίζαμε όμως ε, ήδη τότε ότι δεν θα έφταναν αυτά τα χρήματα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές. Η Τουρκία αναδεικνύεται το ένα και περισσότερο σε παράγοντα κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της γεωγραφικής θέσης, είναι προφανές, αλλά και διότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες ε, στην Τουρκία. Γι' αυτό στα πλαίσια του κοινού σχεδίου δράση ΕΕ Τουρκία για την αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση. Και αναφέρω αυτό το σχέδιο δράση για να έχετε τα συμφραζόμενα. Είναι μια κοινή δράση κατά τη παράνομη μετανάστευση διακίνηση. Ε, ε, ανθρώπων, συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προσφύγων επιτόπου και τις κοινότητες υποδοχής που πρέπει να ε, υποδεχτούν ε, τους ε, πρόσφυγες που καταφθάνουν. Στις 24 Νοεμβρίου συγκροτήθηκε ο συντονιστικός μηχανισμός. Ε, είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο για την Τουρκία και αρχίζει να λειτουργεί από, την, από τον Ιανουάριο του 2016. Τρία δις για το 2016 και 2017. Αυτά αυτό είναι το ποσό ε, της επρικοδότησης ε, του Ταμείου με χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και από τον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δώσουμε τρία δις από τον προϋπολογισμό για τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Θα επανέλθω σε αυτό με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Είναι ένας συντονιστικός μηχανισμός για το ποσό των τριών δις. 500 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό και 2,5 δις από ε, καταλογιστέντα έσοδα από συνεισφορές ε, των κρατών μελών. Είναι, δεν είναι ταμείο λοιπόν, είναι συντονιστικός μηχανισμός. Λοιπόν, είναι εισοδήματα που προέρχονται από τα κράτη-μέλη προς τον προϋπολογισμό για να ενισχυθούν προϋπάρχοντα μέσα, ε, το μέσο για την ανθρωπιστική βοήθεια και το μέσο προενταξιακής ε, βοήθειας, γιατί για την Τουρκία αυτό είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέσο. Οπότε αυτή η φασίλητα, αυτός ο συντονιστικός μηχανισμός επιτρέπει ε, τα κονδύλια να μην διοχετευτούν σε ένα trust fund, αλλά να μπουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης και να ενισχύσουν τα προϋπάρχοντα προγράμματα, διότι θεωρούσαμε ότι αυτό είναι ο απλούστερος τρόπος διοχέτευσης των κονδυλίων, ώστε ταχύτατα να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν γενικότερα για τον προϋπολογισμό, δημοσιονομικός κανονισμός και η υποχρέωση ε, υποβολής εκθέσεων μεταξύ άλλων και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή αυτό ο συντονιστικό μηχανισμό βασίζεται σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δυνάμει του άρθρου 2.10 και 2.14 τη Συνθήκη Λειτουργία τη Ένωση, ε, βάσει τη οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει όποια πρωτοβουλία χρειάζεται για να συντονίσει τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών μέτρων αρρωγή. Ε, και ο στόχο να συντονίσουμε και να ευθυγραμμίσουμε διάφορες επιμέρους δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό της ευρωπαϊκή Ένωσης και από διμερείς συνεισφορές των κρατών μελών, όπως σας είπα. Η μορφή της υποστήριξης ε, είναι ή ε, χορηγίες δάνεια ή άμεση ή έμεση διαχείριση, όπως στη, στη νομική βάση των διαφόρων προγραμμάτων που τώρα εξετάζουμε. Ο συντονισμός θα βασίζεται στην ύπαρξη μια διευθυντική επιτροπή. Steering Committee, παρακαλώ περάστε και στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή η διευθυντική επιτροπή, όπου προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ε, παράσχει στρατηγική ε, κατεύθυνση για... θα εκπροσωπείται φυσικά η Ευρωπαϊκή, Επιτρο... Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβουλευτικό ρόλο θα έχει η Τουρκία μέσα στη Διευθυντική Επιτροπή, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων επιτόπου και όταν κυρίως πρόκειται για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι η αξιολόγηση των αναγκών, η υλοποίηση των δράσεων επιτόπου και ε, ε, η εκτέλεση του σχεδίου δράσης θα γίνεται με συντονισμένο τρόπο και σε καλή συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές, διότι θα αναλάβουν τη διαχείριση των προγραμμάτων. Όπως σας είπα, η όρη η εφαρμοστική είναι η άμεση διαχείριση ή δράσεις για παροχή άμεσης ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Ο στόχος του συντονιστικού μηχανισμού είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων και η υποστήριξη και των κοινοτήτων υποδοχής. Όχι άμεση ε, αρρωγή προς την Τουρκία, προς την τουρκική κυβέρνηση. Θέλω να το τονίσω και αυτό. Οπότε ο στόχος είναι να ε, αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ε, του προσφυγικού, ε, της ροής των προσφύγων και θα υπάρχει ισότητα ε, κατοχυρωμένη ε, ανάμεσα στα δύο φύλλα και ε, μη διακριτική μεταχείριση που θα ηγέται αυτός ο συντονιστικός μηχανισμός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά θα ενημερώνει τακτικά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, τα κονδύλια θα διοχετευτούν μέσω των προϋπαρχόντων προγραμμάτων, οπότε οι αντίστοιχες νομικές βάσεις και εφαρμοστική των προγραμμάτων θα εξακολουθήσουν ε, να εφαρμόζονται, να ισχύουν επιτόπου και ε, οι προθεσμίες επίσης. Ως προς τις ε, εισφορές των κρατών μελών. η προθεσμία είναι 21 Δεκεμβρίου. Παρακαλώ περάστε στην τελική διαφάνεια. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά από τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν πριν από την 21η Δεκεμβρίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή, το χρόνο ε, της, ε, όπου θα καταβάλουν την εισφορά τους και το σχέδιο πληρωμών για ολόκληρο το 2016. Θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πληρωμών. Δεν θέλω να το λέω σχέδιο πληρωμών, πρόγραμμα πληρωμών, να το πούμε, ακούγεται καλύτερο, ούτως να καλυφθούν οι ανάγκες επιτόπου από τις δεσμεύσεις, ε, πρέπει να κάνει την αξιολόγηση επιτόπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι από άλλε συναρμόδιε γαμαδέλτα είναι επιτόπου και κάνουν αυτή την αξιολόγηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα δούμε βάσει του χρονοδιαγράμματο ε, ποιε πληρωμέ θα εκταμιευτούν το 2016 και ποιε θα αναβληθούν για το 2017 ε, σε συνάρτηση με τι ανάγκε. Ε, για να σα ενημερώσω ότι έχει γίνει, χθε, ολόκληρη τη μέρα ήμουνα στην Κορεπέρ, διότι γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο για τι εισφορέ, για το ύψο των εισφορών των κρατών μελών αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, να φτάσουμε τα 500 εκατομμύρια από τον προπολογισμό της Ένωσης ε, και σχεδόν ομόφωνα ζήτησαν τα κράτη-μέλη ε, να είναι υψηλότερο το ποσό που θα βγει από τον προπολογισμό και δεν υπάρχει προφανώς καμία δυνατότητα ε, στον προπολογισμό του 2016, το αναφέρατε κι εσείς, διότι μόλι, ε, πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να ξανανοίξει το προπολογισμό του 2016, διότι όλοι ξέρετε πολύ καλό ότι περιθώριο δεν υπάρχει στο τμήμα 4, όμως θα υπάρχει δυνατότητα ε, να αυξήσουμε την εισφορά από τον προπολογισμό κατά 200 εκατομμύρια το 2017 από το περιθώριο του τμήματος 4 και να κατανομήσει το εσωτερικό του τμήματος αυτού σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει διαθέσιμα ποσά, την διαθέσιμα δηλαδή, κατευθυμισμό γιατί τίποτα δεν είναι διαθέσιμο, ανακατανομή είναι και προσπαθούμε ε, να φροντίσουμε τόσο ότι κανένα από τα προγράμματα που έχει σχέση με την προσφυγική κρίση στις γειτονικές ε, ε, χώρες δεν θα κοπεί, δεν θα διακοπεί για να βρούμε χρήματα για το συντονιστικό μηχανισμό. Ως προς τις φορές των κρατών μελών υπάρχει περιούσα συζήτηση για τη διαχείριση των κονδυλίων και το, για το νομικό πλαίσιο. Στην Κορεπέρ συνεχίζονται οι συζητήσεις και ο στόχος είναι στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξουμε συμφωνία. Οι Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα συμφωνήσουν τις επόμενες ημέρες, οπότε ο συντονιστικός μηχανισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει ήδη από την αρχή του 2016 βλέπετε για το 2016 και 2017 σε αυτό το πίνακα την κατανομή των πληρωμών. Και όπως σας είπα, στην αρχή της παρουσίασης ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, αυτή την ε, πρόκληση και αυτό είναι ένα σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με ποιο τρόπο μπορούμε φιέστερα να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μέσα και βλέπουμε ότι με την κατανομή 2016 και 2017 και τα επιπρόσθετα 200 εκατομμύρια από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας βοηθήσουν να καλύψουμε τις ανάγκες μέσα από αυτά τα μέσα που δεν θέλω να τα ονομάζω ονομάζω δορυφόρους ε, του προϋπολογισμού, διότι θεωρώ ότι προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο το assigned revenue, τα καταλογιστέντα έσοδα, δεν είναι τίποτα καινούριο. Ε, υπάρχουν αυτά στο τμήμα 2, παραδείγματο χάρη, και απλώ το κάνουμε και στο τμήμα 4. Και αυτό μας επιτρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντεπεξερχόμαστε σε... Ε, προκλήσεις ε, που δεν έχουν προβλεφθεί ε, στην αρχικό σχεδιασμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου πριν από δύο-τρία χρόνια. Ήταν πολύ διαφορετικές οι ε, προβλέψεις μας σε σχέση με το μέγεθος, το εύρος της κρίσης που τώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις τις οποίες μας δώσατε. Είναι μια καινοτομία που επηρεάζει τον προϋπολογισμό του 16 που μόλις ψηφίσαμε και γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στον γενικό μας εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επίσης και την δημιουργικότητα και το εφάνταστο των προσπάθειών της για να επιληθεί ένα πρόβλημα στο οποίο ο καθένας θα πρέπει να προσπαθήσει όσο περισσότερο γίνεται για να λυθεί. Είχαμε ένα ταμείο ή ένα καταπίστευμα αν θέλετε για την Συρία με ένα δις 500 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη και 500 από τον προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη όμως δεν σέβονται την υποχρέωσή τους να βάλουν τα χρήματα. Έχουμε ένα καταπίστευμα για την Αφρική, ένα δις 800 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ένα 400 από το Ταμείο Ανάπτυξης και εκεί τα κράτη-μέλη σφυρίζουν κλέφτικα. Και τώρα έχουμε και αυτόν τον καινούριο μηχανισμό που δεν είναι ένα νέο ταμείο, αλλά προσπαθούμε στον μηχανισμό αυτό να του προσδώσουμε ένα κάποιο δεσμευτικό υποχρεωτικό χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη. Ακούγεται λίγο προκλητικό αυτό που λέγω, αλλά ήταν υποχρεωτική η εισαγωγή αυτή. <coughs> το ερώτημα το οποίο τίθεται επίσης είναι το εάν συζητάμε σήμερα για χρήματα τα οποία είχαν καθοριστεί για κάποια άλλα τακτικά ταμεία γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε περάσει να βγάζουμε φωτοτυπίες του χρήματος και να τα διπλασιάζουμε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό εδώ θα μειώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης σε άλλους τομείς. Καταρχάς, ο μηχανισμός αυτός συντονίζεται με το πακέτο για τη μετανάστευση συνολικά με όλους τους άλλους σπόρους, με όλα τα άλλα ταμεία γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένα ταμεία για το ίδιο χοντρικά θέμα. Δεύτερη ερώτηση η οποία τίθεται είναι να δούμε τι επιπτώσεις έχει κάτι τέτοιο στον προϋπολογισμό του 16 γιατί παίρνουμε χρήματα από τον προϋπολογισμό του 16 που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για άλλους ε, λόγους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι απαιτείται περισσότερη ευελιξία και ότι ένας μικρός προϋπολογισμός δεν μπορεί να, ε, να χρησιμοποιείται ε, παντού και πάντα. Πάντως ε, πρέπει να δοθεί μια συλλογική απάντηση σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν θα πρέπει να γίνει αυτό σε επίπεδο διακυβερνητικό αλλά σε επίπεδο κοινοτικό μέσω της κοινοτικής μεθόδου. Τι σημαίνει αυτό για τον προϋπολογισμό του 16, 500 εκατομμύρια, εντάξει. Το θέμα είναι όχι τι θα κάνουμε με τα 500 εκατομμύρια που θα πάρουμε, αλλά τι δεν θα κάνουμε με τα 500 εκατομμύρια τα οποία θα βγάλουμε από τον προϋπολογισμό. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε τον τρόπο μέσω του οποίου θα εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την διαδικασία. Θα υπάρξει ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός, υποτίθεται, θα υπάρξουν συμπληρωματικοί πόροι στον προϋπολογισμό, πόροι οι οποίοι μπαίνουν στον προϋπολογισμό χωρίς να μπουν ουσιαστικά, χωρίς να υπάρχει προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Όλα αυτά ακούγονται περίεργα, δεν ξέρω πώς θα γίνουν. και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αγαστά ε, με το ε, Συμβούλιο και με τα άλλα όργανα. Και τέλος θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα καταστήσουμε τις χώρες πραγματικά υπεύθυνε και υπόλογες στις επιλογές τους. Ε, με τα trust funds, με τα καταπιστεύματα το πράγμα δεν πήγε καλά. Αυτός ο μηχανισμός προβλέπεται κάπως πιο περιοριστικός Ελπίζω να υπάρξουν κάποιες αποδοτικές επιτέλους συζητήσεις στο Συμβούλιο. Επανειλημμένα έχω πει εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι το θέμα της αλληλεγγύης δεν είναι θέμα διακηρυκτικό. Το να βγάζεις ανακοινώσει δεν είναι αλληλεγγύη. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα περάσουν στην πράξη για να δείξουν εκεί με ποιο τρόπο είναι αλληλέγγυα. Να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπα και στην αρχή, τεράστια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφάνταστη πρακτική που ακολούθησε για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται πάρα πολύ να το ελέγξουν. Και ως εισηγητής του 16 εκφράζω την αλληλεγγύη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ έτσι ώστε η Επιτροπή μας, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να συνεχίσουν να πιέζουν έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και να επιληθεί επιτέλους ένα τέτοιο σημαντικότατο πρόβλημα. Ευχαριστώ, Χριστοφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συμφωνήσω με όλα όσα ανέφερε ο συνάδελφο ο κ. Φερνάντε. Θα πω ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο, 145 τόσα δι. Δεν πιστεύω να υπάρχει πουθενά σε κανέναν εχειρίδιο οικονομική θεωρία που θα λέει ότι όταν ορίζεται ένα προπολογισμό, αυτό ο προπολογισμό ορίζεται με την υποσημείωση ότι θα καλύψει και οποιασδήποτε άλλε έκτακτε ανάγκε προκύψουν. Πιστεύω ότι αυτό ανατρέπει τα πάντα Πάβει να εφίσταται σαν προπολογισμό όταν αυτέ οι έκτακτε ανάγκε ποτέ δεν προπολογίζονται και είναι ένα άγνωστο σχή. Άρα, όπω απαγορεύεται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν ελλείμματα, έπρεπε να απαγορεύεται να καλύπτονται από τον προπολογισμό οποιασδήποτε έκτακτε ανάγκε. Έπρεπε να υπάρχει τρόπο, επιτέλου πρέπει να διαδραματίσει πιθανό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που το παίζει ανεξάρτητη, ως αν και να μην συνδέεται και αυτή με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λέω για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέλος, εάν αφαιρούμε και αυτές τις έκτακτες ανάγκες, είτε προσφυγικό λέγεται, είτε οτιδήποτε άλλο, από τον προπολογισμό, οι πολίτες και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού κάθε χρόνο θα μειώνεται ο προπολογισμό και οι δυνατότητες του, δεν θα έχουν λόγο να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η τακτική θα οδηγήσει τελικά και στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν την επόμενη χρονιά το προσφυγικό απαιτεί 30 δισεκατομμύρια θα διαλύσει ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διαλύοντας τον προπολογισμό θα διαλυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλοι πρέπει να συνδράμουν και να βρουν τρόπους και λύσεις. Πιστεύω ότι έπρεπε να δημιουργηθεί άλλο ταμείο για έκτακτες ανάγκες από άλλους πόρους με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πιθανώς και άλλους και βάσει αυτού να κινείται να καλύψει τι οποιασδήποτε έκτακτε ανάγκε. Επί του προκειμένου όσον αφορά το ζήτημα με την προσφυγικό. Ο κύριο Ντούσκ χθε εμά μα είπε ότι δώσαμε 18 δισεκατομμύρια γενικά για τα ανθρωπιστικά και το προσφυγικό. Θα ήθελα να γνωρίζω και εδώ πρέπει να γίνει και ενημέρωση. Δώσαμε 18 δις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στημένη στον τοίχο και την πυροβολούν γιατί δεν κάνει τίποτα για το προσφυγικό. Θέλω να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στοιχεία τι έδωσαν τα αραβικά κράτη, τι έδωσαν που αν τα αραβικά κράτη δίνανε ένα πετροδολάριο το βαρέλι, πιθανώς να εκάλυψαν το πρόβλημα όσον αφορά την οικονομική πτυχή. Τι έδωσαν οι άλλες χώρες, οι άλλοι οργανισμοί δεν ξέρω πώς φτάσαμε να θεωρείται αποκλειστικά θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το προσφυγικό. Δηλαδή αυτέ οι χώρε 28 που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτέ ανήκει το προσφυγικό. Οι άλλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη ούτε για το οικονομικό, ούτε για την επανεισδοχή, ούτε για την αντιμετώπιση των ροών. Αναφέρατε ότι η Τουρκία είναι κλειδί. Κανένα δεν αφισβητά τον ρόλο τη Τουρκία. Δεν τη θεωρώ ότι είναι το κλειδί γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, το πρόβλημα αν θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτή την υποστήριξη θα έπρεπε να την δώσουμε στον πρώτο σταθμό που κάνουν οι πρόσφυγες, που είναι ο Λίβανος και η Ορδανία, που έχουν πολύ περισσότερους πρόσφυγες, που η οικονομία τους είναι πολύ πιο αδυνατή από την Τουρκία, δεν αντέχουν και δεν σηκώνουν που αν σπάσει αυτή η δυνατότητα από τον Λίβανο και την Ιορδανία, πιστεύω θα είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα από ότι είναι με την Τουρκία. δεν συμφώνησαν οι χώρε να δώσουν τα 2,5 δι και πρέπει να μα το επιβεβαιώσετε. Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω μια χώρα που δεν θα δώσει ούτε έναν ευρώ γιατί θεωρείται ανύπαρκτη από την Τουρκία. Αυτή η χώρα είναι δική μου, η Κύπρο. Όταν αναφέρεται η Τουρκία και ο Γλου αναφέρεται σε μια νήσο που είναι τυχαία στη Μεσόγειο και δεν υπάρχει ούτε ονοματολογία ούτε αναγνωρίζει την ύπαρξη. Άρα σίγουρα δεν θα αναγνωρίζονται και τα λεφτά μα. Δεν θα τα δώσουμε, δεν θα δώσουμε μία ούτε ένα ευρώ. Άλλωστε η Τουρκία αν ήθελε να πάρει λεφτά από την Κύπρο θα έπαιρνε πολύ πιο εύκολα αποσύροντα το στρατό που τη κοστίζει μερικέ εκατοντάδε εκατομμύρια το χρόνο και τον έχει εκεί να τον κρατά η ευρωπαϊκή χώρα. Άρα από την Κύπρο δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι δεδηλωμένη και δεδομένη θέση μα. Άρα μια χώρα δεν θα συνεισφέρει προ την Τουρκία και για αυτόν τον λόγο και για πολλού άλλου. Η ανησυχία μου θα πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει μέσω τη Τουρκία. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε Κούρδοι που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στο Κοπάνι και στη Συρία. Και η Τουρκία του κρατεί σαν πρόσφυγε και δεν του επιτρέπει να πάνε στο Κοπάνι πίσω γιατί φοβάται τη δημιουργία κουρδικού κράτου και την ενίσχυση των Κούρδων γιατί θέλουν, θέλει να επικρατήσουν οι Τουρκμένοι μέσα στη Συρία. Δηλαδή παίζει παιχνίδι με του πρόσφυγε ακόμα και με αυτού που θέλουν να πάνε πίσω στη Συρία. Έχει δεκάδε χιλιάδε. Εμένα μου είπαν ότι είναι εξακόσε χιλιάδες. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι λιγότεροι. Δεν του επιτρέπει, έκλεισε τα σύνορα και δεν του αφήνει και του κρατάει στην Τουρκία. Θα χρηματοδοτούμε και αυτού του πρόσφυγε που του κρατάει η Τουρκία με το έτσι θέλω, με τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτά πιστεύω είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή πιθανώ και το Συμβούλιο. Και ε, ένα τελευταίο ε, αν δοθούν αυτά τα λεφτά τα τρία δις ε, πρέπει να βρεθεί και ένας μηχανισμός να ενημερωνόμαστε πού πάνε αυτά τα λεφτά κάθε αν όντως πάει και το τελευταίο ευρώ πραγματικά στους πρόσφυγες ή χάνονται με αυτά τα κόλπα που θα επινοήσει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι γνωστός τακτικιστής. Θεωρώ ότι τελικά να συμφωνήσω με την Επιτροπή. Είναι κλειδί η Τουρκία γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία είναι μέρος του προβλήματος η Τουρκία είναι αυτή που έχει μεγάλη συμβολή στο να φτάσουμε ενό εδώ και να δημιουργηθεί το προσφυγικό με την τακτική που εφάρμοσε στην γύρω περιοχή. Και θα συστήσω προσοχή όταν έχετε να κάνετε διαχείριση με την Τουρκία. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Χριστοφόρου. Βεβαίως η διερμηνία διακόπτη στι 12.30 και έχω ακόμα και γραμμένα μέλη. Κύριε Γκούρινς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάφορα σχόλια. Πρώτον, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του θέματος και διευκρίνηση ορισμένων πτυχών. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι τα χρήματα που θα διατεθούν στην Τουρκία δεν θα περάσουν από τα ταμεία του τουρκικού κράτους, θα πάνε σε οργανισμούς οι οποίοι θα προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Για τη χρηματοδότηση έχω το εξή σχόλιο. Από χρόνια τώρα ζητούμε πρόσθετα κονδύλια. Ο ανθρωπιστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών είναι χρόνια υποχρηματοδοτούμενος. Αυτό έχει γίνει πια διαρθρωτικό χαρακτηριστικό και όχι συγκυριακό. Τρίτο, Και εδώ θα συμφωνήσω με τον Γενικό Εισηγητή. Μέχρι τώρα πληρώνουμε συμβολικά ποσά για την ελάφρυνση των συνθήκων στα στρατόπεδα του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Τώρα, το καταπιστεύω, το Trust Fund. Οι χώρες ζητούν 1,8 δις. Είμαστε περίπου στο 5% του ποσού που ζητείτε. Άρα Είμαστε πιο κοντά σε ένα ε, ε, προϊόν το οποίο ανακοινώνεται αλλά ποτέ δεν έρχεται παρά στην πραγματικότητα. Πάλι και αυτό πάει να γίνει συστηματικό. Οι χώρες μέλη ζητούν, υπόσχονται μέσα στο 0,7% εδώ και δεκαετίες ήμουνα και στη διάσκεψη του Μοντρέ και της Αντισανταβέβα που έχει προβλέψει νέους στόχους που υποτίθεται ότι θα πληρωθούν με το 2015, μετά γίνεται πάλι αναβολή. Άρα οι χώρες μέλη υπολείπονται των υπεσχημένων και για τα trust fund για την Αφρική και για τα όσα υπόσχονται εν προκειμένου. Θα έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα στα χέρια μας. Όλοι οι ανθρωπιστικοί φορείς αναμένουν τι θα ανακοινωθεί, μάλλον αυτά που θα ανακοινωθούν να υλοποιηθούν κιόλας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, θα, θα οδηγηθούμε σε αναπρογραμματισμό. Αναπρογραμματισμό υπό διάφορους τίτλους. Μη λησμονείτε ότι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν πρώτα υποστήριξη ανάπτυξης. Τέλος, δηλαδή πάρουμε από αλλού κονδύλια για να διαθέσουμε εκεί. Και σημειώνεται μια γενική τάση απογύμνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα προνομιά του. Εδώ χρειάζεται ταχύτατη δράση και αποφασιστική στο στάδιο αυτό για να επιληθεί πρώτα, να, να προσπαθήσουμε να, ε, ε, να επιλύσουμε πρώτα το πρόβλημα των εξουσιών του Κοινοβουλίου, αυτό το κάνουμε στη διαδικασία της ε, αναθεώρησης, όταν θα πλησιάζουμε και όλα στο 2020. Διότι σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως, το Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο. Όσον αφορά το καταπίστευμα, το Trust Fund για τα χρήματα που έρχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, πάλι το Κοινοβούλιο δεν έχει τίποτε άλλο, απλώς ενημερώνεται. Σε ό,τι αφορά τούτο εδώ το Ταμείο, πάλι εδώ είναι εντελώς περιθωριακή η εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Θα χρειαστεί να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό είναι ο μακροπρόθεσμο στόχο. Για το βραχυπρόθεσμο στόχο να έλθουν οι χώρε μέλη να εξηγήσουν και εδώ, ενώπιον μα, τι γίνεται. Χρειάζεται ένα σύστημα το οποίο να αναγκάζει τι χώρε μέλη να υλοποιούν τα υπεσχημένα. Να έλθουν να εξηγήσουν γιατί δεν φτάνουν μέχρι το 0,7%, γιατί προβαίνουν σε ανακοινώσει αλλά μετά δεν τηρούν τα υπεσχημένα. Πρέπει να λεχθεί καθαρά Ποιο είναι υπεύθυνο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η διακυβερνητική ε, ε, προσέγγιση η οποία τελικώ ευθύνεται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι αρχηγοί καθών και κυβερνήσεων αναλαμβάνουν τώρα και ε, δεσμεύσει για την COP21. Ναι, ναι, πρόκειται για μασκαρά τα κανονική, λέει ο κ. Γκέρνης. Αυτή είναι ωστόσο η εικονική πραγματικότητα, α το πω έτσι. Ολμπριχτ. Ένα σύντομο σημείο για τον προϋπολογισμό. 0,5 του προϋπολογισμού θα πρέπει να αναπρογραμματιστεί στο κεφάλαιο 4. Ε, προκαθορισμένα εξωτερικά έσοδα. Τι σημαίνει αυτό για τα 2,5 δις. Σημαίνει ότι θα έχουμε επιπλέον 2,5 δις τα οποία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό και αυτή τη στιγμή ενταχθούν στον προϋπολογισμό πού θα πάνε. Θα πάνε και αυτά στο κεφάλαιο 4 ή υπάρχει κάτι το ε, πιο συγκεκριμένο στον προϋπολογισμό. Ποιος είναι εν πάση περιπτώσει ο μηχανισμός κατανομής θα είναι επιπλέον τα χρήματα αυτά. Ίσως ο κύριος Φερνάντες να μας το εξηγήσει αυτό σε, με δημοσιονομικούς όρους. Ποιος είναι ο μηχανισμός και πού είναι τα χρήματα. <laughs> Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέει ο Πρόεδρος, να μας πει. Να εκδώσει και να κόψει καινούριο χρήμα. Βάνα. Έχω και εγώ ερωτήσεις όπως οι προηγούμενοι ομιλητές για το ποσοστό συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Προϋπολισμού και των χωρών μελών. Υπάρχει μία έγγραφο από χθε του Συμβουλίου που λέει ότι θα επιβαρύνουν και τα 3 δισεκατομμύρια τον ευρωπαϊκό προπολισμό και ότι δεν προβλέπεται συνεισφορά των χωρών μελών. Μήπως υπάρχει κάποια παρανόηση εδώ. Στο μη έγγραφο δεύτερο, επί του περιεχομένου, κάποιος το είπε και πριν, για το περιεχόμενο των μέτρων, η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για το ποια μέτρα θα πρέπει να προβλεφθούν, είναι αρκετά σαφές. Αφενός μιλεί για ανθρωπιστικά μέτρα υπέρ των προσφύγων, έχει καλώς, μετά όμως μιλεί γενικά για μέτρα στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την διαχείριση του προσφυγικού. Εδώ χωράνε πολλές ερμηνείες. Η ερώτησή μου είναι, περιλαμβάνονται εδώ και αστυνομικά μέτρα, μέτρα προστασίας των συνόρων, θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτούν και τέτοια, ή εδώ αποκλείεται κάποια μέτρα. Κύριε Συναδινέ. Ευχαριστώ πολύ εκπλήσωμαι από την ταχύτητα αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ενίσχυση της Τουρκίας. Σας έχει καταλάβει αμικός ο φόβος του Ισλαμικού κινδύνου που για χρόνια ένας από αυτούς που εκτρέφει τον Ισλαμικό κίνδυνο είναι η Τουρκία και εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο στέλνοντας μετανάστες πρόσφυγες προς τη γυραιά Ήπειρο προσπαθείτε να πείσετε τους εαυτούς σας όλοι ότι εάν προσφέρετε τη βοήθεια των τριών δις στην Τουρκία θα μειωθεί ο κίνδυνος. Πλανάστε πλάνη νικτράν. Διότι ιστορικά και διαχρονικά η Τουρκία δεν σέβεται καμία απόφαση μεγάλου οργανισμού δεν σέβεται επί χρόνια τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών όσο αφορά το Κυπριακό. Κατέχει το 1 τρίτο του νησιού και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της αυτές τις αποφάσεις και έχετε την εντύπωση ότι θα σεβαστεί το φόβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισδοχή των μεταναστών στο έδαφος της Ευρώπης. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ήδη έχει δοθεί στην Τουρκία το κονδύλιο των 130 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη μεταναστών κατά την περίοδο 11-13. Έχουν σχεδιαστεί άλλα 245 εκατομμύρια για την περίοδο 14-16. Επιπλέον έχει κινητοποιηθεί βοήθεια ύψους 94 εκατομμυρίων για τον ίδιο λόγο. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εισέρχεται κύμα μεταναστών από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Μάλλον η Κομισιόν εκτιμά ότι τα παραπάνω κονδύλια που δόθηκαν είναι λίγα για την Τουρκία και θέλει να τις δώσει επιπλέον τρία δις. Ρωτώ λοιπόν, στην περίπτωση που η Τουρκία λάβει τα κονδύλια, αλλά οι μετανάστες δεν μειωθούν, σκοπεύει να δώσει και άλλα χρήματα ή θα επιβάλλει κυρώσει στην Τουρκία διότι δεν μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους της. Πώς θα εξασφαλίσει η θα επιβαλλει κυρωσεις στην τουρκια διοτι δεν Ένωση ότι τα κονδύλια που θα δώσει στην Τουρκία θα διατεθούν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή το να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές ή θα χρηματοδοτηθούν άλλοι τομείς. Εάν δεν συνεισφέρουν όπως σχεδιάζεται κράτη-μέλη για τη συγκέντρωση του ποσού των 2,5 δις, πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα κονδύλια. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να πιστεύει ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με όσα ανέφερα παραπάνω. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη. Δεν θα ήθελα εδώ να ασχοληθώ με το πολιτικό κομμάτι του θέματος, το ποιος πήρε την απόφαση αυτή. Βέβαια αυτός θα έπρεπε να αναλάβει και την ευθύνη. Το θέμα είναι το έλεγχος του ταμείου αυτού. Βρισκόμαστε σε μια κατεπίγουσα κατάσταση και είδαμε ότι σε τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις θα έλεγα ο έλεγχος είναι συνήθως ανεπαρκής Ακριβώς γιατί τα χρήματα δίδονται πάρα πολύ γρήγορα και οι συνθήκες ελέγχου είναι περιορισμένες. Θα ήθελα λοιπόν, εφόσον βρεθούν τα χρήματα αυτά, θα έχετε ένα σύστημα για να τα ελέγξετε σε μια χώρα σαν την Τουρκία και θα δείτε με κάποιο τρόπο τα χρήματα αυτά να φτάνουν στον στόχο τους γιατί αλλιώς θα ήταν άχρηστη η προσπάθεια. Μέχρι τώρα οι ερωτήσεις που έχω θέσει δεν έχουν αποδώσει καθόλου. Μαραγκάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει, η οποία προσπαθεί από το τίποτα να βρει μια λύση. και το παρουσιάζει το θέμα σαν να ήταν κάτι το φυσιολογικό, το κανονικό, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι κατά της ιδέας αυτής, ίσα ίσα είμαι υπέρ. Αλλά για να είναι κανείς υπέρ θα πρέπει να έχει ε, έναν σαφέστατο προσανατολισμό για τη συνεισφορά των προπολογισμού από πλευρά των κρατών μελών και για τον προορισμό των ποσών αυτών. Αν κάτι τέτοιο, ε, αν, θα έλεγα κάτι χρειάζεται μια σαφέστατη δημοσιονομική δομή, αυτό είναι. Αυτά τα 2,5 εκατομμύρια από τα δις από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα κριθεί να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, υπάρχει αναγκαιότητα θα έλεγα, να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και για τα έσοδα και για τον προορισμό των ποσών αυτών. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι ε, στην ουσία ομολογούμε όλοι την πλήρη τεράστια άγνοιά μας ε, γύρω από τα θέματα. Τι θέλουμε να καλύψουμε, ποιες ανθρωπιστικές ανάγκες ε, θέλουμε ε, να καλύψουμε. Ξέρουμε χοντρικά πού θέλουμε να πάνε τα λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα πάνε εκεί που θέλουμε. Θα θέλαμε λοιπόν με το μέσο αυτό να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε με πολύ υπευθυνότερο τρόπο. Το πρόγραμμα λοιπόν μας ενδιαφέρει αλλά πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τη διαχείριση του προγράμματος. Αυτό είναι υποχρέωσή μας. Εκτιμώ, επαναλαμβάνω, την προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι για την αποσία του Συμβουλίου που ασχολείται με την αναθεώρηση την ενδιάμεση του MFF. Αλλά όπως είπε ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει να μιλάμε για μια ιονή δημοσιονομική πολιτική σε σχέση με τέτοια θέματα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για κανονικές ε, ε, συνθήκες συναλλαγής με μια χώρα η οποία είναι χρήσιμη, φίλη, συνεργάζεται. Ε, εδώ με την Τουρκία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η λογική λέει ας δώσουμε τα χρήματα για να μην έρθουν όλοι αυτοί εδώ. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είμαστε απλά καχύποπτοι, είμαστε ανήσυχοι σε σχέση με το θέμα αυτό. Απέναντι λοιπόν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Τουρκίας πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και επιφυλακτικοί. Και θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να μπορούσαν να είναι πολύ πιο δραστήρια στην υποδοχή των προσφύγων δεν πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε και ιδιαίτερα την κατάσταση στις χώρες προέλευσης. Merci. Σας ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την δεκάλεπτη παράταση που μας έδωσαν. Θα ήθελα, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Καλβίνιο, να διευκρινίσω κάτι. Αυτός ο προπολογισμό εντάσσεται τελικά στον προπολογισμό τη Ένωση. είναι κάτι ξεχωριστό. Δεύτερον, κυρία Καλβίνιο, οι δεσμεύσει που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη για το Αφρικανικό και το Συριακό ε, Ταμείο ε, πώς έχουν πρικοδοτηθεί και ποια είναι η κλίδα κατανομής. Έχει αποφασιστεί ή ε, ο καθένας ε, κάτω δοκούν θα συνεισφέρει. Λοιπόν, είναι 12.30, έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Και υπάρχουν και δύσκολες πολιτικά ερωτήσεις. Όταν ε, όμως υπάρχει πυρκαγιά δεν κάθεται κανείς να συζητήσει πόσο κάνει το νερό τη ημερών ημέρα. Για να αναχαιτήσουμε ε, τις προσφυγικές δροές ε, ε, αυτό, από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία και από τον πόλεμο και έρχονται στην Ευρώπη. Ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά εύστοχα όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα ήθελα αρχίζοντας να σας πω πως συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα σχόλιά σας. Πρέπει να είμαστε ε, σε επαγρύπνηση, πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί για τη χρήση των κονδυλίων που στόχο έχουν να ε, ανταποκριθούμε σε αυτή τη μαζική ροή προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρέσα για να σχολιάσει τα τεχνικά ζητήματα για τον προϋπολογισμό, αλλά θα ήθελα να ε, σας καθησυχάσω, κύριε Όλμπριχτε, τα, δεν ακουμπάμε τα υπόλοιπα trust funds. Ε, τις επιστώσεις θα τις πάρουμε από τα top-up των προγραμμάτων που συμφωνήσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2016. Και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο γιατί μέχρι τελευταία στιγμή επέμεινε Αυτά τα προγράμματα, συγκεκριμένα το ΕΠΑ και το ENI, να ενισχυθούν. Ε, και αυτό έγινε στη τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Τα ποσά υπάρχουν ήδη στον προϋπολογισμό και στην νομική βάση προβλεπόταν ότι θα διοικητευτούν ε, στην ε, ε, Τουρκία και έχουμε και το, την, το εφεδρικό για την ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα ποσά υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό του 2016. Και ο κύριος Χριστοφόρου έθεσε επιτάπητος ένα ε, πολύ σημαντικό στοιχείο ε, ότι δίνουμε την εντύπωση ότι παραμένουμε αδρανείς, δεν κάνουμε τίποτα. Νυχθημερών εργαζόμαστε. Η Επίτροπος Γεωργίευα ήθελε να έρθει, αλλά δεν μπορούσε να έρθει διότι πήγε στην Ελλάδα ε, για την υπογραφή συμφωνίας με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Όλοι καταβάλουν πραγματικά μέγιστες προσπάθειες ε, για τα κονδύλια του προϋπολογισμού έχουν διπλασιαστεί τα ποσά. Παρ' όλα αυτά επικρατεί η εντύπωση ότι επιτόπου δεν κάνουμε αρκετά. Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα πηγαίνει μέσω μη κυβερνητικών και άλλων διεθνών οργανισμών ε, στο στόχο τους και τα ποσά του τμήματος 3 είναι αντικείμενο μικτής διαχείρισης ε, με τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν λόγω της μαζικής ροής να απορροφήσουν πλήρως αυτά τα ποσά. Και κάποια μέσα που ε, έχουν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ε, θα χρησιμοποιηθούν, αλλά παίρνουμε χρήματα από το ΑΜΙΦ για τους πρόσφυγες ε, και από το ESF, από το Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχουν πάντως όντως από πλευράς κρατών μελών αδυναμίες ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων. Ακούσαμε διάφορα ερωτήματα σε σχέση με το, το, στόχο ε, που ακριβώς θα διοχετευτούν τα κονδύλια. Συνάδελφοι από την Κύπρο και από την Ελλάδα αναρωτιούνται αν τελικά τα χρήματα δεν θα καταλήξουν στην Τουρκία. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο στόχος αρρωγή προς τους μετανα... πρόσφυγες και προς την ε, κοινότητα υποδοχής Δηλαδή δεν θα μπουν στον προϋπολογισμό της Τουρκίας αυτά τα χρήματα. Τι μέτρα, κοιτάξτε, το, το πρώτο κύμα είναι παραδοσιακή ανθρωπιστική βοήθεια. Ερυθρός Σταυρός, ε, τη αρμοστία ε, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ε, διάφορες δράσεις. Σα είπα ότι γίνεται αξιολόγηση των αναγκών αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και τις άλλου οργανισμού του ΙΕ και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και φαίνεται να συμφωνούν μαζί μα. Δηλαδή το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν είναι σε προσφυγικού καταβλισμού και είναι εκτό και μάλιστα στι φτωχότερε περιοχέ τη Τουρκία είναι ξεκάθαρε όμω οι ανάγκε και εντοπισμένες ε, ε, ε η βοήθεια, ε, ε, υπηρεσίες υγείας, ε, βασική εκπαίδευση για τα παιδιά, ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά. Αυτή είναι η άμεση υποστήριξη και στη συνέχεια πρέπει να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες υποδομές για την παροχή αυτών των υπηρεσιών ε, κέντρα, ε, πρωτογενής ε, περίθαλψη και ούτω καθεξής και ανάπτυξη κατόπιν της υποδομής. Η αξιολόγηση των αναγκών ξεκάθαρα επικεντρώνεται στους πρόσφυγες και στις κοινότητες ε, υποδοχής. Και το καταλαβαίνω ότι ανησυχεί το Κοινοβούλιο, θα ανησυχούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπαίνουν τα χρήματα στον προϋπολογισμό ε, της ε, Τουρκίας. Συνεχίζεται αυτή η άσκηση αξιολόγηση και θα σας κρατούμε ενήμερους όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, για την αίρεση τώρα, για τη χρήση των κονδυλίων, σας είπα ότι ε, υπάρχει το στρατηγικό κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ Τουρκίας και εκεί εντάσσεται ο συντονιστικός μηχανισμός και υπό αίρεση φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια από τις τουρκικές αρχές και σας είπα ότι δεν είναι ένα καταποκοπή ποσό που θα μεταφερθεί κάπου. Όχι, θα υπάρχει μια συνέχεια πληρωμών σύν το χρόνο για να καλύπτουμε τις ανάγκες σταδιακά θα εκταμιεύονται τα ποσά. Σας είπα θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το 2016 και 2017 και θα τα παρακολουθεί τις πληρωμές η Διευθυντική Επιτροπή Steering Committee για να κατοχυρωθεί η πτυχή αυτή από την, ε, για τις πληρωμές. Ε, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη πως πέρα από τα ευρωπαϊκά μέσα. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται πάρα πολύ και είναι εξαιρετικά γενναιόδωρα σε διμερές επίπεδο και δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Όταν μιλάμε για τις δράσεις των κρατών μελών, νομίζω είναι πιο δίκαιο να το αναφέρουμε. Κυρία Βένα, ρωτήσατε ε, τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το έγγραφο ε, που κυκλοφόρησε στο Συμβούλιο, ότι τα, τα τρία δις ε, θα βγουν από τον προϋπολογισμό. Κυκλοφόρησαν αυτό το τεχνικό έγγραφο, η Γερμανία και η Γαλλία, η Κόρεπερ δεν ενέκρινε αυτό το τεχνικό έγγραφο. Γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και περιμένουμε να λάβουμε μηνύματα στα τηλέφωνά μας. Προς το παρόν απόφαση δεν υπάρχει, ούτε και πρόταση εναλλακτική από πλευρά του Συμβουλίου. Μια στιγμή να δω τις σημειώσεις. Ερεσιμότητα. Τέλος, για την ταχύτητα δράσεως και ορισμένες ανησυχίες για αυτό το fast engagement. Τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός αποτελεί όργανο ή εργαλείο που για ορισμένους ίσως δεν είναι επαρκές για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά έχει ορισμένα στοιχεία ευελιξίας που μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε σε ορισμένες προκλήσεις, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Πέρσι είδαμε, για παράδειγμα, την κρίση στην Ελλάδα, που ήταν ε, το θέμα που απασχολούσε πάρα πολύ Ιούνιο και Ιούλιο. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός έδωσε έξτρα 2 δισεκατομμύρια πληρωμές το 2015 και 2016 με μεταφορά πιστώσεων μέσα στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Ταχύτατη αντίδραση για να αντιμετωπιστεί μια επίγουσα κατάσταση. Μετά, η ε, κρίση των γαλακτοπαραγωγικών. Άλλη κρίση αυτή αντιμετωπίστηκε με 700 εκατομμύρια. Τώρα αντιμετωπίζουμε άλλη κρίση. Νομίζω ότι είναι ω σωστό να αναγνωρίσει κανεί ότι υπάρχουν και ορισμένα θετικά στοιχεία. Το γεγονό δηλαδή ότι μπορούμε να βρούμε ευφύς τρόπους, δημιουργικούς τρόπους είπε κάποιο πριν, για να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε και να αναζητήσουμε λύσει μέσα στο νομικό πλαίσιο που διαθέτουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου καθώς και πολιτικής λογοδοσίας εξακολουθούν να ισχύουν όπως είναι η περίπτωση και σε τούτην εδώ την διευκόλυνση facility βρίσκοντας λοιπόν αυτές τις ευφυείς λύσεις στην ουσία τελικά αυτό μας πληρώνεται να κάνουμε. Άρα υπάρχει ένα θετικό μήνυμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε προς τα έξω και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και καλύτερα με, τον, με το κοινό και δράση επιτόπου είναι αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε και βεβαίω αυτό που θέλουν πρωτίστως οι πρόσφυγες επιτόπου. Μου επιτρέπετε να περάσω το μικρόφωνο στον Σιλβάνο για να σας εξηγήσει πώ λειτουργεί ο μηχανισμό διαθέσεως των πιστώσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα 2,5 δις έξτρα χρήματα που προστίθενται στο μισό ε, ε δις του προϋπολισμού, πώς θα λειτουργήσουν αυτά. προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επιτρέπει δηλαδή δοτές εκτός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να συνεισφέρουν σε συγκεκριμένα εργαλεία, ιδίως για την ε, εξωτερική βοήθεια, να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν δηλαδή στην εφαρμογή. Θα αυξηθούν λοιπόν έτσι τα χρήματα που είναι διατεθειμένα, που είναι διαθέσιμα μάλλον, για ένα συγκεκριμένο σκοπό, είτε για ανθρωπιστική βοήθεια, είτε το λεγόμενο προενταξιακό εργαλείο. Και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει περισσότερα μέσα τότε για την εφαρμογή των πολιτικών της και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το συγκεκριμένο στόχο για την ενίσχυση των προσφύγων στην Τουρκία. Αυτό δεν αποτελεί τύπης μέρος των ε, ε, πιστώσεων του ετήσιου προϋπολογισμού, αλλά τα κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα το 2016 και 2017 θα προσθεθούν σε αυτά δηλαδή τα 2,5 δις σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα. κάποιος διακόπτει, διακόπτει ο πρόεδρος Με συγχωρείτε κύριε Ρεζά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ειδικό μέσον ή θα είναι ο ίδιος ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ο προϋπολογισμός της Ενώσεως και είναι συγκεκριμένα κονδύλια, συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού που εξουσιοδοτούν για την δαπάνη και καθορίζουν ποια είναι τα επιλέξιμα κονδύλια και ποιες είναι οι επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και μέσω του προενταξιακού εργαλείου. Εκεί καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα ίδια ισχύουν και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και εδώ ε, τίθεται και το θέμα των ελέγχων. Ρώτησε ο κ. Βάλλη ποιο ελέγχει. Αφού η εφαρμογή γίνεται μέσω των εργαλείων του προϋπολισμού, όλοι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται τώρα θα εφαρμόζονται. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μειώνεται το επίπεδο ελέγχου. Θα ελέγχονται πλήρως ε, οι δαπάνες που, στο οποίο ο προϋπολογισμός. Άρα για τον προϋπολογισμό 2016 θα εγγραφεί ένα δις 500 εκατομμύρια έξτρα εσόδων. Δηλαδή το μισό των 2,5 δισεκατομμυρίων που υποτίθεται θα συμβάλλουν οι χώρες μέλη το 2017. Ο κύριος Ρεζά. Δεν είναι εγγεγραμμένα η διαθεσιμότητα για το 2016 των ε, μέσων για τις δράσεις υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία θα αυξηθούν κατά το ποσόν αυτό, κατά το τμήμα αυτό των εξωτερικών συνεισφορών που δεν χρειάζονται εξουσιοδότηση από την αρχή επί του προϋπολογισμού αφού πρόκειται για ατομικές συνεισφορές των χωρών μελών. Εμφανίζονται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Είναι έσοδα που θα μπουν στις δράσεις του προϋπολογισμού. Ναι, άρα λοιπόν 1,5 δισεκατομμύριο αλλά αυτό θα επιτρέψει να αυξηθεί κατά 1,250 δις ε, τα μέσα για την προένταξη και τα διάφορες γραμμές του προπολισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα Ποια θα είναι η κατανομή στις χώρες. Η πρόταση της Επιτροπής είναι η κατανομή των βαρών να βασιστεί στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα που είναι ο κανόνας του προϋπολογισμού και είναι βέβαια οικείος ο τρόπος αυτός υπολογισμού για όλες τις χώρες μέλη. Άρα το μόνο που λείπει είναι η έγκριση των χρονομερών. Χε, χε, χε. Αλλά είμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ίσως αυτό να βοηθήσει. Και ε, μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε. Τελειώσαμε. Ε, θυμήστε μας τι μένει ακόμα για τα Trans Fund ε, Αφρικής και Συρίας. Πόσο. Ένα δις, ένα δις 200 εκατομμύρια. Προτιμώ να σας απαντήσω γραπτός για να σας δώσω και πιο επίκαιρα νούμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευκρινήσεις, ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε ως τώρα και ευχαριστώ και τους μεταφραστάς. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα, αντιπροσωπεία δηλαδή, θα μεταβεί στην Τουρκία από 8 έως 10 προσεχούς Φεβρουαρίου. Και με την ευκαιρία αυτή θα καταστεί δυνατόν να δούμε πώς οργανώνεται αυτή η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Ούτως ή άλλως ώστε να μείνουν μάλλον στην Τουρκία και να μην έλθουν στην Ευρώπη. Έχετε άλλες ερωτήσεις. Δεν πειράζει αν δεν έχετε. Η επόμενη συνάντησή μας θα διεξαχθεί του χρόνου στις Βρυξέλλες 27 και 28 πρώτου. Στο μεταξύ σας εύχομαι καλές γιορτές. Σε όλους και όλους.